Ah, Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε. Πριν να ξεκινήσουμε τις ε, εργασίες μας, ε, θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Γιάννος Λαββαλέζα, ε, είχε ένα πολύ κακό οδικό ατύχημα ε, και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο αλλά δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πάντως, ως πρόεδρος της Επιτροπής μας ε, έστειλα άμεσα ένα μήνυμα με ευχές εξ ονόματος της Επιτροπής μας, ευχόμενη βεβαίως ταχύ ανανάρρωση και ε, θα ε, λαμβάνω νέα για την πορεία αποκατάσταση υγείας του Αδέλφου και θα σας μεταφέρω τα νέα αυτά. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας ε, είναι η έγκριση του σχεδίου ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρείται εγκεκριμένη. Επόμενο σημείο, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων για τις συνεδριάσεις της 14ης-15ης Ιουνίου και της 12ης και 13ης Ιουλίου του 2011. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα και τα πρακτικά αυτά. Α, πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις εργασίες των συντονιστών. Στη διάρκεια των, της συνάντησης των συντονιστών, λοιπόν, συζητήσαμε πρώτα απ' όλα την οργάνωση ε, ερευνητικών αποστολών. Τον Ιούλιο ήδη είχαμε ε, συζητήσει και αποφασίσει για τον Οκτώβριο ε, να οργανώσουμε δύο αποστολές, μία στο Βερολίνο και μία στη Ρουμανία η Γραμματεία είχε αρχίσει να εργάζεται για την προετοιμασία αυτών των, των αποστολών, αλλά δημιουργήθηκε κάποια προβλήματα όσον αφορά τον... την παρουσία ε, το... αυτών με τους οποίους θέλουμε να συναντηθούμε ε, στις συγκεκριμένες χώρες και επομένως απεφασίστη να μετακινηθούν λίγο οι ημερομηνίε και να οργανωθούν οι δύο αυτές αποστολές στις 24 και 25 Νοεμβρίου ταυτοχρόνως το προσχέδιο των εργασιών των αποστολών θα σας διανεμηθούν ως ο νούπο μέσα στις επόμενες ημέρες μαζί με την σύνθεση των αποστολών. Επιβεβαιώνεται επίσης το πρόγραμμα για το επόμενο έτος, το πρόγραμμα των εργασιών όπου θα επισκεφθούμε τις χώρες που δεν καταφέραμε να επισκεφθούμε στη διάρκεια του 2011, κυρίως δε τη Γαλλία, την Ιταλία, την Γερμανία, ε, στα όρια με την ε, Τσεχική Δημοκρατία καθώς και την Πολωνία εγκρίναμε το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Επιτροπής μας για το 2012 ε, υπό την αίρεση των δύο ε, ε, συνεδριάσεων το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο που έχουν προβληθεί ταυτόχρονα με άλλες επιτροπές συγκεκριμένα με την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων ε, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα και σε μένα και σε άλλα μέλη της Επιτροπής θα αποφασίσουμε τι θα γίνει στην επόμενη ε, φορά που θα συναντηθούμε διανεμήθη το πρόγραμμα το οποίο μάλλον είναι οριστικό, το πρόγραμμα του σεμιναρίου της 6ης Οκτωβρίου και που αποφασίσαμε να οργανώσουμε μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα συζήτηση για την εφαρμογή των ε, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μοιράστηκαν επίσης στους συντονιστές, μάλλον εδόθησαν στους συντονιστές κάποιες ανακοινώσεις από πλευράς επιτρόπων και άλλων θεσμικών οργάνων ε, όσον αφορά ανοιχτές και υποσυζήτηση αναφορές. Έχουμε επίσης λάβει πρόσκληση από τον Ευρωπαίο Μεσολαβητή για να συμμετάσχουμε δι' αντιπροσώπων μας ε, στο 8ο σεμινάριο των Μεσολαβητών 21 και 22 Οκτωβρίου του 2011 στην Κοπενχάγη και αποφασίσαμε να απαντήσουμε ζητώντας από τους συναδέλφους Όκεν και Ιτουργκάης να συμμετάσχουν σε το εν λόγω σεμινάριο εκπροσωπώντας την Επιτροπή μας. Επίσης, Επίσης επιβεβαιώθηκε η παρουσία ε, του Επιτρόπου Ποτότσνικ στις εργασίες της Επιτροπής μας ε, τον μήνα Νοέμβριο ενεκρίθη, ε, δόθη δηλαδή μια πρώτη έγκριση στο άτυπο προσχέδιο ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Δεν είχαμε άλλες ανακοινώσεις και επομένως Ολοκληρώθηκε και η ανακοίνωση της Προέδρου σχετικά με τις εργασίες των συντονιστών και περνούμε επομένως στο επόμενο σημείο που είναι οι εργασίες της σήμερα μεταξύ των κεντρικών ε, σημείων μας στο 8 ε, υπάρχει μία αναφορά σχετικά με τη διατήρηση της καφέ αρκούδας στην Γαλλία ε, που θα παρουσιάσει ο κύριος Φρανσουά Αρκάντζελη. Στο σημείο 13 επίσης μία αναφορά σχετικά με τους συμβασιούχους υπαλλήλους στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφορά η οποία θα συζητηθεί παρουσία των αναφέρομεν, των, του αναφέροντος μάλλον. Θα έχουμε επίσης ανταλλαγή απόψεων και μία πρώτη συζήτηση στην την έκθεση Ρουγκάη σχετικά με τα απόβλητα και θα συνεχιστεί η συζήτηση για την έκθεση Nord Stream. Αυτά για σήμερα. Έχουμε επίσης ε, ένα κατάλογο με τις συστάσεις ε, σχετικά με τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί σε κάποιες ε, αναφορές. Εάν οι προτάσεις αυτές σας βρίσκουν σύμφωνους, τότε θα συμπεριληφθούν στις επόμενες συνεδριάσεις. Υπενθυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε ολομέλεια στο Στρασβούργο. Την Τρίτη το απόγευμα θα έχουμε συζήτηση για την, έκθεση, για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής μας. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να είναι παρόντες έτσι ώστε ε, να στηρίξουν την εισηγήτρια Μάγερ. Και στο τέλος, ε, μετά το πέρας της συζήτησης στην Ολομέλεια, θα οργανώσουμε μια, μια συνέντευξη τύπου, όπως κάναμε και πέρσι, γιατί μετά από μια πρώτη ε, έτσι, ε, μετά από μια πρώτη μάλλον ε, συζήτηση είδαμε ότι θα πρέπει να στείλουμε τελικά και ένα έγγραφο σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως. Πρώτη αναφορά λοιπόν που έχει εγγραφεί που αφορά το περιβάλλον είναι αναφορά που έχει υποβάλει ο κύριος Παναγιώτης Μπούρας, ελληνικής ηθαγένειας, εξ του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεγαλόπολης σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρου των ελληνικών αρχών, κοινοτικών κριτηρίων και διαδικασιών υποδοχή των αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευή χώρου υγειονομική ταφής αποβλήτων κοντά στην πόλη Μεγαλόπολη, ε, στην περιφέρεια της Πελοποννήσου στην Ελλάδα. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον και επομένως θα δώσω αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας διέφυγε το όνομα, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά αυτό το σχέδιο στην, ε, αυτό το, στην Μεγαλόπολη, να υπενθυμίσω ότι τη 10η Σεπτεμβρίου 2009 κατεδικάστη η Ελλάδα ε, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή ε, κοινοτικών κριτηρίων καθώς επίσης και για την ελληπή εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για την υγειονομική ταφή αποβλήτων θα πρέπει ε, να έπρεπε οι, ελληνικές ε, αρχές λαμβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές ε, οδηγίες να έχουν δημιουργήσει το εν λόγω δίκτυο. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγαλόπολης δεν έχει ε, λάβει γνώση το, της ε, μελέτης ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη. Επομένως, ακόμα τα πράγματα είναι εξαιρετικά ασαφή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο? Μποστινάρου. It is an déjà vu We must... Έχουμε την αίσθηση ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό το σκηνικό. Θα πρέπει να σταματήσει. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δίνει καμία απάντηση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ε, αν είναι αρμόδιες. Καμία απάντηση από τις τοπικές αρχές. Νομίζω ότι όταν συζητάμε την έκθεση για το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ε, τα χρονικά περιθώρια και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την απάντηση ε, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι το μοναδικό, το μοναδικό συμπέρασμα που μπορούμε να εξαγάγουμε γιατί οι αρχές δεν ε, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για όσα συμβαίνουν στους πολίτες και θα πρέπει να σταματήσει η κατάσταση αυτή. Άλλες ε, παρεμβάσεις ο Γιάννη. Ε, Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι συχνά δεν λαμβάνουμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Γίνεται μια σχετική μελέτη περιβαλλοντική συμβατότητας. Βρίσκεται και στην παρούσα φάση υποανάπτυξη, θα την εξετάσουμε και μετά θα κοιτάξουμε τα αποτελέσματα. Αλλά για τους αναφέροντες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τι νόημα έχει, θεωρούν, να γίνονται όλες αυτές τις διαδικασίες, αν σε δύο χρόνια γνωρίζουμε ότι τα πράγματα θα έχουν πάει λάθος. Θα πρέπει να καλέσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τα κρατημέλη προκειμένου να χορηγούν τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της περίπτωσης. Γιατί θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι όποιο δεν χορηγεί τα σχετικά στοιχεία ε, είναι ένοχος. Γιατί αν φτάσουμε και ξέρουμε εκ των πραγμάτων ότι έχει γίνει λάθος, θα είναι πλέον πάρα πολύ αργά. Θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά γιατί δεν έχουμε ακόμα οριστικά αποτελέσματα αλλά παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει την Ελλάδα να χορηγήσει τα σχετικά στοιχεία. Σαλαβράκος. Κύριε Σαλαβράκο. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα την απάντηση της Επιτροπής. Ε, δεν αλλάζει τίποτα από την απάντηση που μας είχε δώσει στις 20 Φεβρουαρίου του 2009. Όμως εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου του 2011 φέτος ε, μια κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα την έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων για το έργο το υποσυζήτηση. Ε, θα παρακαλούσα λοιπόν να μείνει ανοιχτή μεν η αίτηση του Δημάρχου, η αναφορά του Δημάρχου, αλλά ε, ο παριστάμενος ο πρόσωπος ε, της Επιτροπής να ζητήσει άμεσα να λάβει γνώση των νέων στοιχείων και να συζητηθεί η υπόθεση μέσα στον χρόνο διότι η Ελλάδα από καθυστερήσεις τέτοιου είδους υφίσταται πρόστιμα. Και ναι μεν δέχομαι ότι πρέπει να εξετεστούν όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τις επιδράσεις τους των αναφέροντες, αλλά παράλληλα δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και να λέμε ότι από τη μια βάζουμε πρόστιμα στην Ελλάδα και από την άλλη ε, δεν μεριμνούμε τουλάχιστον να έχουμε τις εξελίξεις της ελληνικής πολιτείας πάνω στο θέμα. Παρακαλώ λοιπόν τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να λάβει ε, τα στοιχεία αυτά τα οποία θα τα δώσω εγώ είμαι πρόθυμος να το δώσω και να έρθει η υπόθεση πάλι εντός του έτους παρακαλώ. Να μην πάμε σε καινούριο χρόνο και έχουμε καινούρια πρόστιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Επομένως αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά. Ε, και βεβαίως κάνοντας έκκληση για μία ακόμα φορά στην Επιτροπή όσον αφορά και την ουσία αλλά και όσον αφορά και την μεθοδολογία βέβαια και την το χρονοδιάγραμμα ε, ε, να σέβεται λοιπόν και το χρονοδιάγραμμα, μια και εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έχει ζητηθεί ήδη επανειλημμένα. Περνάω στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Είναι αυτό που έχει εγγραφεί στο σημείο 7. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τη οδηγία για διαχείριση των αποβλήτων βάσει των αναφορών που έχουν ληφθεί. Η συγητής ε, είναι ο συνάδελφος στον οποίο θα δώσω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα στην παρουσίαση αυτής της έκθεσης για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στα κράτη-μέλη και σχετικά με, ε, το θέμα του, των αποβλήτων γενικότερα, θα ήθελα να αναφερθώ στις πολιτικές ομάδες και να τις ευχαριστήσω διότι με βοήθησαν και μπόρεσα να ανταποκριθώ στο έργο μου γιατί χρειάστηκε να κάνουμε πολλές συνεδριάσεις πρόεδρε για να φτάσουμε σε έναν καλύτερο προγραμματισμό αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα τα οποία οδηγεί σε πληθώρα αναφορών. Πρόκειται για το ότι οι δημόσιες αρχές δεν μπορούν ικανοποιητικά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει πολλά νομοθετικά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει μια πλαισίωση, μια νομική πλαισίωση, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο σύγχρονο τρόπο ζωής μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα απόβλητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των βιομηχανιών, των νοσοκομείων, των σπιτιών μας και των γραφείων μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθούμε. Διαφορετικά υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για την υγεία αλλά και για την βιωσιμότητα του πλανήτη. Κρίνοντας από τις αναφορές βλέπουμε ότι η ανησυχία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος πολλών κοινοτήτων. Δηλαδή βλέπουμε ότι το θέμα μετατρέπεται σε ένα πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα και οι πολίτες περιμένουν από εμάς να εγκρίνουμε αυτή την νομοθεσία. Άρα αυτό που διακυβεύεται είναι η αξιοπιστία της ε, κοινοτικής νομοθεσίας. Γι' αυτό με αυτή την έκθεση προσπάθησα να λύσω προβλήματα τα οποία έχουν θέσει και οι αναφέροντες. έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα της ε, διαχείρισης των αποβλήτων. Έχει σημασία να ευαισθητοποιήσουμε και τους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας μιλήσω για συμπεράσματα αυτής της έκθεσης για να δούμε τι θα γίνει με την διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, θα ήθελα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία πλαίσιο περί αποβλήτων με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης των αποβλήτων. Επίσης, να αναγνωρίσουμε ότι δεν γίνονται αρκετές επενδύσεις για έργα υποδομής και διαχείρισης των αποβλήτων στα περισσότερα κράτη-μέλη και επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα ταμεία σύνοχης, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν ορισμένα σχέδια και προγράμματα. Το ίδιο αφορά και την ΕΤΕ. Επίσης, ε, ως προς υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτό το τομέα, θα πρέπει να έχουν μια σωστή κατάρτιση. Το γραφείο μας, ο Οργανισμός Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, επίσης, θα μπορούσε να συντονίσει καλύτερα τα κράτη-μέλη για να δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν και να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταποκριθούν στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης, χρειάζεται μια καλύτερη στρατηγική διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί απασχόληση και έσοδα. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για μια πιο αποδοτική διαχείριση αποβλήτων. Έκτον, θα πρέπει να γίνει σωστή εφαρμογή της οδηγίας για την αξιολόγηση επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος μέσα στα πλαίσια της αδειοδότησης που προβλέπει η κάθε εθνική νομοθεσία. Έβδομον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επαγρυπνούν έτσι ώστε να γίνει σωστή μελέτη αντικτύπων πριν ε, γίνεται η εγκατάσταση μίας, ναι, μάλλον πριν από μία νέα εγκατάσταση ε, διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης, ο διάλογος μεταξύ δημοσίων αρχών, ο ιδιωτικός τομέας και η συζήτηση με τον πληττόμενο πληθυσμό είναι ο καλύτερος τρόπος για να ορίσουμε τις προτεραιότητες για την στρατηγική, την διαχείριση και τη στρατηγική μας για την αντιμετώπιση των αποβλήτων. Ένατο, ζητάμε από την Κομισιόν να προτείνει σαφέστερα κριτήρια έτσι ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις για τους επικείμενους κινδύνους στην ανθρώπινη, για την ανθρώπινη υγεία. Και επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της επικουρικότητας. Άρα θα πρέπει να εντάσσονται όλα αυτά τα στοιχεία στο κοινοτικό δίκαιο, ιδιαίτερα ως προς τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας για την αποτίμηση των κινδύνων επί του περιβάλλοντος και να δούμε κατά πόσο υπάρχει πραγματική προστασία της φύσης και της ιστορικής κληρονομιάς. Γι' αυτό χρειάζεται ένας ορισμός ως προς τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων, καθώς και ένα σύστημα παρακολούθησης, παρακολούθησής τους. Επίσης να υπάρχουν κυρώσεις καθώς και αποτρεπτικά μέτρα για τις παράνομες απορρίψεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τοξικές ουσίες, για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το περιβάλλον και, εν πάση περιπτώσει, ο πάντα να πληρώνει. Αυτά τα σημεία και όλα όσα βλέπετε στην έκθεση, στην ουσία θέλουν να επαυξήσουν αυτές τις ανάγκες, αυτή την ανάγκη, δηλαδή ότι αυτή η έκθεση αποτελεί απαράβατο όρο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, αφού είδαμε σωρία αναφορών που συνεχίζει να υφίσταται και τώρα για τα απόβλητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών μας, να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση, να δεχτούμε και τις τροπολογίες και στη συνέχεια να συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια. Νομίζω θα γίνει αυτό το Δεκέμβριο. Και ελπίζω να φτάσουμε σε μία έκθεση αυτής μας της Επιτροπής η οποία να περιλαμβάνει όλες τις επικρίσεις και τις ανάγκες που μας αναφέρουν τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι αναφέρονται Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Συνάδελφε Ιντουργκάης για την ε, εργασία την οποία ε, έχετε εκπονήσει θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χειροντίας Δεκαστήλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Um, I work at, um, unit. Είμαι στην ε, υπηρεσία C2, στη μονάδα C2 για, την, ε, για θέματα αποβλήτων. Εξετάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το σχέδιο της έκθεσης. Η έκθεση όντως ε, ε, θέτει μερικά ερωτήματα, τα οποία, ζητήματα τα οποία τα γνωρίζουμε σωστά, καλά, για την σωστή ε, διαχείριση των αποβλήτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία για, την, για τα απόβλητα αλλά και για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δυστυχώς υπάρχει, συνεχίζεται να σπαταλάτε αυτό το θέμα των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τάση για ανακύκλωση και λιγότερη υγειονομική ταφή. Αλλά Όταν λέμε ανακύκλωση, εννοούμε ανακύκλωση σύμφωνα με τα καλύτερα δυνατά πρότυπα, σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές τεχνικές. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει μια πολύ αντιφατική, αν θέλετε, και μια εικόνα με πολλές αντιθέσεις από Χώρε σε χώρα. 16 χώρες ε, προβαίνουν σε υγειονομική ταφή μεγαλύτερου ποσοστού του 50% των ε, ε, αποβλήτων. Οι, οι έξι που δεν το κάνουν αυτό είναι οι συνήθεις υποπτή. Η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία και έχουμε πέντε χώρες, ε, την Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, που έχουν, αν θέλετε, ένα μείγμα διαχείρισης αποβλήτων. Προβαίνουν σε κάυσες κυρίως, σε λιγότερες υγειονομικές ταφές και ε, λίγη ανακύκλωση. Αυτή την κατάσταση αντιμετωπίζουμε λοιπόν και πάνω από το 20% όλων των παραβιάσεων ε, που έχουν να κάνουν με θέματα περιβάλλοντος αφορούν τα απόβλητα. Άρα μου φαίνεται πολύ κέρδο το γεγονός ότι τίθεται το θέμα αυτό. Αλλά εξ όσων καταλαβαίνουμε σε πολλές καταγγελίε πολιτών χρησιμοποιούνται πάρα πολλοί πόροι από πλευρά ε, επιτροπή και Κοινοβουλίου και κανείς το καταλαβαίνουμε αυτό δεν θέλει να ζει δίπλα σε χιτά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι όσο παράγουμε απόβλητα θα χρειαζόμαστε τέτοιους χώρους. Φυσικά όλοι αυτοί οι χώροι θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα. Επίσης, να σημειώσω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αναφέροντες απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πρώτη αρχή και παρά το γεγονός ότι ασκούν ένα δικαίωμά τους, θα έπρεπε πρώτα να απευθυνθούν στις τοπικές, εθνικές αρχές και μόνο στη συνέχεια δεν υπάρχει σωστή ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές αρχές. Επίσης, ξέρω ότι αυτό απασχολεί πολλούς, ε, πολλές αναφορές. Όταν φτάνουν σε μας ε, οι αναφορές, το project, τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ε, χορηγηθεί ακόμα σχετικές εγκρίσεις και άδειε. Αυτό αφορά κυρίως τη δημιουργία χώρων ταφής και καύσεως. Και πάλι αυτό, αυτό απασχολεί ιδιαίτερα τους, το κοινωνικό περίγυρο, τους κατοίκους της περιοχής, αλλά Δυστυχώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την νομική αρμοδιότητα στη φάση εκείνη να διαπιστώσει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άρα δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου πραγματοποιηθεί το έργο για να παρέμβουμε. Να ολοκληρώσω τώρα αναφέροντας ποιες είναι οι προτεραιότητές μας σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα απόβλητα. Ήμουν ε, επί 3,5 χρόνια υπεύθυνο για την οδηγία για του ΧΙΤΑ και καταλαβαίνω λοιπόν τι προβλήματα προκύπτουν και σε ό,τι αφορά την οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά. Θα πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο του 2010, από ό,τι ξέρετε, έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, δεν έχουμε καθόλου καλές ε, καλά στοιχεία σχετικά με την μεταφορά. Άρα αυτό θα πρέπει να το θέσουμε στο επίκεντρο των προσπάθειών μας, προκειμένου να παίζουν όλα τα κρατημέλη με τους ίδιους κανόνες. Και αν θέλουμε να έχουμε τη σωστή επίλυση ενός προβλήματος, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε τα σωστά στοιχεία. Θα πρέπει να περάσουμε πέρα από το επίπεδο της ε, Eurostat και να συλλέξουμε πιο πολλές πληροφορίες. Χρειαζόμαστε την ε, βοήθεια υπηρεσιών όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, όπως ανέφερε προηγουμένως ο κ. Ιτουργκάης. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, στοιχεία που να στέκουν. Επίσης θα πρέπει να ελέγξουμε την εξωτερική εφαρμογή της οδηγίας πλαίσια για τα απόβλητα και θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας. Τα ευρωπαϊκά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και κάθε φορά όταν λέω αυτή τη λέξη μου έρχεται στο νου η καμπανία γιατί όπως ξέρετε στα χαρτιά όλα ήταν τέλεια αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα και τώρα αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα στην καμπανία. Τα γνωρίζει λοιπόν τα προβλήματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει στενά να παρακαλουθήσει τι γίνεται στις χώρες που δεν βρίσκονται, ας το πούμε έτσι, στην κορυφή των μέτρων για τη διαχείριση αποβλήτων. Αυτές οι 16 χώρες που ανέφερα. Αλλά και τα προγράμματα πρόληψης ε, δημιουργίας αποβλήτων και αυτά θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί μέχρι το 2013 και ξέρετε δεν είναι νωρίς να αρχίσουμε να ασκούμε πιέσεις στα κρατημέλη για την προετοιμασία των προγραμμάτων αυτών. Όπως είπα, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν μηχανισμοί για να πληρωθούν τα κενά που έχουμε ως προς τα στοιχεία μας, ως προς τις γνώσεις μας και θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους διάφορους οργανισμούς, τα διάφορα θεσμικά όργανα. Βρισκόμαστε σε συνεργασία και με τον Ευρωπαϊκό ε, Οργανισμό Περιβάλλοντος. Θα συνεχίσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να βοηθά τα κράτη-μέλη μέσω καθοδήγησης, μέσω υποστήριξης να κατανοήσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μου φαίνεται ότι η στάση της Επιτροπής είναι αμφιλεγόμενη γιατί από τη μία πλευρά καλεί, οθεί τους ε, πολίτες ε, για πιο συμμετοχικές διαδικασίες και από την άλλη πλευρά εδώ ε, συμβουλεύει τους ιδίους ε, πολίτες πρώτα να περιμένουν ε, να εξαντλήσουν όλα τα εθνικά μέτρα και εθνικές αρχές πριν στραφούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα τότε σε πολλές περιπτώσεις όπως και στην περίπτωση της καμπανίας που εσείς αναφέρατε τότε τα πράγματα έχουν ήδη, τα, προβλήματα έχουν ήδη παγιωθεί και είναι ακόμα πιο δύσκολη η λύση. Εγώ εν τω μεταξύ θα δώσω τον λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Συνάδελφος Μέρκης πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον αγαπητό συνάδελφο για την εκτενή παρουσίαση της εργασίας σας και ευχαριστώ και την αγαπητή της Επιτροπής. Το θέμα των αποβλήτων είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη και για την Επιτροπή μας ε, και πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί μια απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και, ε, όσον την αντιμετώπιση του προβλήματος και βεβαίως είναι σαφές και αυτονόητο ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι. Και αυτό υπογραμμίζεται στην έκθεση. Απ' την άλλη πλευρά, όσο καλό είναι, τόσο ασαφές είναι. Γιατί είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να γίνεται ε, σεβαστός ο νόμος και η νομοθεσία. Γιατί πρέπει να το ξαναλέμε τι να σας πω, η Επιτροπή Αναφορών ε, θα πρέπει να υπογραμμίζει την ανάγκη ε, τήρησης της νομοθεσίας στην Ευρώπη, δεν νομίζω. Αντιθέτως, νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε μια απάντηση σε όλους αυτούς τους αναφέροντες που φτάνουν μέχρι εμάς. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ζητήσω από τον εισηγητή η έκθεση, η αυτή, η έκθεση του να μην είναι αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς είμαστε ένα νομοθετικό σώμα, δεν ε, ε, είμαστε εδώ απλώς για να ζητούμε κάποια πράγματα. Επομένως, σε αυτήν την σημαντική έκθεση θα πρέπει ε, να δίνουμε απαντήσεις στους αναφέροντες. Και επίσης θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχουμε μία σταθερή πορεία. Δηλαδή κάθε φορά που ε, λαμβάνουμε ε, εκθέσεις θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τρόπο αντιμετώπισης των αναφορών ε, εάν ε, το μέγεθος αναφοράς είναι α ή β ή εάν η σημασία, η σοβαρότητα του θέματος είναι ε, τέτοια και εν πάση περιπτώσει να ξέρουμε αν πρέπει να ζητήσουμε την διαδικασία επί παραβάση ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι θα πρέπει πάντως να έχουμε ένα είδος format, ένα είδος τυποποιημένων I think... Ένα είδος τυποποιημένων απαντήσεων λοιπόν. Γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα φτάσουμε στην καρδιά του ζητήματος. Γιατί λοιπόν υπάρχουν τόσες πολλές αναφορές, ε, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, γιατί, δεν, γιατί υπάρχει ελλειπής δράσης όσον αφορά ε, τα θέματα αυτά, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα θέματα αυτά και ε, ε, γιατί οι πολίτες μας δεν θέλουν ας πούμε να υπάρχει ένας ε, information and they are indeed not ε, ένας αποτεφρωτής στην πίσω τους αυλή ή δύο βήματα από το σπίτι τους νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να βρεθούν λύσεις γιατί ε, οι πολίτες μας ε, πραγματικά ε, απασχολούνται από τα θέματα αυτά. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι μόνο η έλλειψη των πόρων ένα κομμάτι των, ε, της εφαρμογής της νομοθεσίας θα πρέπει να το αναλαμβάνουν οι εθνικές ε, κυβερνήσεις. Ε, δεν είναι δυνατόν πάντα να στρέφονται προς εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε να ξεφορτωθούν ας πούμε τα απόβλητά τους. I, therefore, do not think that we should turn Επίσης, ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να στρεφόμαστε πάντα προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Νομίζω ότι η στροφή προς, τις, προς τα διαφορετικά ταμεία ε, είναι μια ενδιάμεση λύση και ελπίζω ότι θα αποτελέσει ενδιάμεση λύση και για την ε, καμπάνια. όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να συζητηθούν και με το περιβάλλον και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, να κάνουμε ε, κάποια κοινά αιτήματα κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν όμως κατά την άποψή μου και κάποια μέτρα που μπορεί να έχουν ταχύτερη ε, θετική επιρροή. Ας πούμε, αυτό που είδαμε στην Ιταλία ε, είναι ότι υπάρχει μια ατελείωτη σειρά, ατελείωτος αριθμός υπαλλήλων που υποτίθεται ότι ε, πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα αλλά δεν ασχολούνται αποτελεσματικά. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε ποιοι και πώς ε, ασχολούνται, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι και πώς ασχολούνται με το θέμα αυτό. Επίσης θα πρέπει να αρχίσει να ασχολείται με το θέμα, να την προσκαλέσουμε κιόλας την υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος να αποκτήσει μια νέα εντολή ενδεχομένως αυτή ε, η υπηρεσία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι δεν έχουμε τη σωστή νομοθεσία, αλλά πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η νομοθεσία αυτή και πώς εφαρμόζεται. Άρα ε, χρειάζεται διαφάνεια και η διαφάνεια θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σημεία της έκθεσής σας. Επικίνδυνα απόβλητα. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίε. δεν έχουμε πάρα πολλές αναφορές συγγνώμη, για το θέμα αυτό. Ενδεχομένως θα αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον. Πάντως δεν πιστεύω ότι η αποτέφρωση των ε, επικινδύνων αποβλήτων είναι ε, το, το αυτή καθεαυτή πολύ ε, σημαντικό πρόβλημα. Η, έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη διαβούλευσης με τους πολίτες, αυτά είναι τα σημαντικά προβλήματα. Αγαπητέ συνάδελφε ε, και αγαπητοί συνάδελφοι γενικώ, νομίζω ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι σημαντικό και στο μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι τα απόβλητα ε, θα αποτελέσουν πηγή ενέργειας για το μέλλον. Η ανακύκλωση θα μας δώσει νέες πρώτες ύλες για το μέλλον και επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις αναφορές αυτές και με έναν τρόπο διαφορετικό να τις αντιστρέψουμε έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα αυτά στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρτίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος διότι με κάλυψε συνάδελφος Μέρκης. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Ιτουργκάης γιατί νομίζω ότι η έκθεσή του είναι χρήσιμη και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Είναι μια σοβαρή έκθεση, διότι πολλές φορές δεν υπάρχουν όρια ή προδιαγραφές εργασίας. Καταρχήν, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προτεραιότητές μας. Και πιστεύω ότι αυτή θα πρέπει να είναι μία από τις λίγες εκθέσεις που επιβάλλεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια με τις νέες διαδικασίες που υπάρχουν. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί υπήρξε ομοφωνία. Αλλά πολλές φορές ψηφίζουμε χωρίς να γίνει καν παρουσίαση. Επειδή είναι κάτι που είναι ύψης της σημασίας, θα έπρεπε να συζητηθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της έκθεσης και να την πάμε στην Ολομέλεια, ζητώντας να γίνει μια εκτενή συζήτηση. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το ότι θέτει ορισμένα όρια για να προσπαθήσουμε να εξορθολογήσουμε και την εργασία της δικής μας της Επιτροπής σε ένα πολύ σημαντικό τομέα που καταφέρνει να φτάσει σε μία σχετική πλειοψηφία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια και η κυρία Μέρκης έχει απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να εντάξουμε αυτόν τον τρόπο εργασίας όχι ως πλατφόρμα αναζωπήρωσης διαφόρων, αλλά επίλυσης προβλημάτων. Και σε σχέση με αυτά που είπε η Ουδίφ, είπε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές σε αυτό το τομέα γιατί υπάρχει ευαισθητοποίηση. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλές αναφορές διότι δυστυχώς γίνεται μεγάλη μόλυνση. Δεν υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση ως προς το θέμα της μόλυνσης. Βεβαίως έχουμε προχωρήσει και σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπεται να δίνει, δεν επιτρέπεται τα σούπερ μάρκετ να δίνουν πλαστικές σακούλες, αλλά παρόλα αυτά ε, γίνονται, γίνεται μόλυνση, μόλυνση τεραστίων διαστάσεων. Πολλές φορές πρέπει να εξηγούμε και στα μικρά παιδιά τι συμβαίνει, δηλαδή να μην ξεχνάμε ότι όποιος μολύνει, μολύνει ολόκληρη την κοινωνία και θα πρέπει οι πολίτες να ξέρουν ότι φέρουν ευκρινή δεν, μπορούμε δηλαδή να μιλάμε για τα απόβλητα και για τη σωρία αποβλήτων τη στιγμή που τα δημιουργούμε εμείς πρώτοι-πρώτοι. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε, να συγχαρώ και τον Κάρλος και θα δούμε, Πρόεδρε, κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε με τα θέματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ πολύ, ο Σάνσβος Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, εισηγητή γιατί τα κατάφερε πάρα πολύ καλά σε μια πολύ δύσκολη ε, σε ένα πολύ δύσκολο έργο να βάλει ένα σύστημα και να κάνει μια πολιτική δήλωση για το πρόβλημα αυτό. Και έτσι μπορεί όχι μόνο να ψηφιστεί από την Ολομέλεια, αλλά να συζητηθεί και όλο αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά η έκθεση αξίζει να συζητηθεί. Μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Το φαινόμενο αυτό το έθιξε φυσικά και η κυρία Μερκής. Γιατί σε κανονικές συνθήκες τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Καταρτίζουμε νομοθεσία και περιμένουμε από τα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν. Αλλά εμείς ποιο φαινόμενο αντιμετωπίζουμε ότι συχνά δεν συμβαίνει αυτό η δάλος, δεν θα λαμβάναμε αναφορές και έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα, όταν καταρτίζουμε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν προθεσμίες και αυτό φυσικά είναι εύλογο. Οι χώρες άλλωστε χρειάζονται χρόνο μέχρι ότου εφαρμόσουν την νομοθεσία, αλλά σε αυτή την μεταβατική περίοδο, όταν λαμβάνουμε μία αναφορά και την ε, θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει «Μα γιατί ενίσταστε» εφόσον υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος. Και μετά περνάει αυτή η μεταβατική περίοδος και διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Άρα χρειάζεται, θεωρώ, και μία παρακολούθηση, να μην φτάνουν η μέρα της ε, λήξης της προστασμίας και να μην έχουμε κάνει τίποτε. Και η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη σε ό,τι αφορά τα απόβλητα. Γιατί τα απόβλητα στις πιο πολλές χώρες αποτελούν θέμα τοπικής αρμοδιότητας. Δεν είναι της ε, κεντρική κυβέρνησης. Σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μακριά από εμά δηλαδή, το επίπεδο αντιμετώπιση των ε, αποβλήτων. Και σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και μια ιστορία πίσω από κάθε πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό είναι η έλλειψη πληροφοριών, η έλλειψη στοιχείων. Το ακούσαμε και αυτό σήμερα. όταν έχουμε μπροστά μας μία αναφορά και μας γίνονται καταγγελίες και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει τι απαραίτητε πληροφορίε, αυτό είναι παράδεκτο. Δεν είναι το ελάχιστο το οποίο χρειαζόμαστε όταν μα περιγράφεται μια κατάσταση από τα... έναν αναφέροντα και ζητάμε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει η Επιτροπή να λαμβάνει τι πληροφορίε που χρειάζονται. Γιατί πολύ συχνά ο τοπικό βουλευτή, ο εθνικό βουλευτή γνωρίζει την κατάσταση πολύ πιο καλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, ε, παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας αλλά και καλύτερη διαβίβαση των πληροφοριών. Και εμείς χρειαζόμαστε πιο πολλές πληροφορίες γιατί το περιβάλλον ανήκει σε όλους μας. Το πρόβλημα των αποβλήτων είναι εγκάρσιο και με εγκάρσιο τρόπο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και Γκίτο, ε, ανέλαβες βαρύ έργο, αλλά πραγματικά χαίρομαι που τα πήγε τόσο καλά. Και το ξαναλέω ότι θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να μην διεκπαιρεωθεί μόνο αυτή η έκθεση στην Ελλομέλεια αλλά να συζητηθεί κιόλα. Ευχαριστώ πολύ, ο την Άρου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ιτουργκάη, τον αντιπρόεδρό μας και να τον συγχαρούμε θα ήθελα όμως να δούμε ποιες θα είναι οι πρακτικές συνέπειες αυτής της έκθεσης, διότι θα είναι ένα μέσον για να αλλάξουμε την τρέχουσα κατάσταση, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Μιλήσαμε για τη Μεγαλόπολη και είδαμε ότι δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το θέμα εμείς ως μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα σε επίπεδο οργανισμών και ιδιαίτερα περιφαλλοντικών οργανισμών. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται επίσημη διαβούλευση όταν μιλάμε για διαχείριση αποβλήτων. Πήγαμε στη Βουλγαρία και είδαμε ποια είναι η γραφειοκρατία και πολλές φορές αποκλείονται και από την αίθουσα εκείνοι οι οποίοι προβάλλουν καλά σχέδια, ενδιαφέροντα σχέδια. Και δεν είμαστε μόνοι εμείς οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι. Επίσης, άρα δεν υπάρχει σωστή διαβούλευση. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί σωστά μία μελέτη επιπτώσεων, μελέτη αντικτύπου. Πώς γίνεται η αξιολόγησή τους, διότι τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που οδηγούν σε μεγάλο αριθμό αποβλήτων και τοξικών ουσιών ε, ιδιαίτερα επικινδύνων, θα πρέπει να τονίσουμε, κύριε Ιτουργκάης, ότι θα πρέπει να ορίσουμε νέες αρμοδιότητες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ε, κινδύνους πριν γίνει η αξιολόγηση. Δηλαδή να μην δεχόμαστε τις θέσεις των κυβερνήσεων και των οικονομικών φορέων και των κυβερνήσεων πολλές φορές ε, προβάλλουν μια συμπεγνία με τους οικονομικούς οργανισμούς. Επίσης, να ορίσουμε τον χρόνο αντίδρασης για τις εθνικές κυβερνήσεις, τους τοπικούς φορούς, φορείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στην περίπτωση της ε, ε, Μεγαλόπολης δεν απαντάν οι τοπικές αρχές ούτε η εθνική κυβέρνηση και άρα έρχεται η Κομισιόν και μας λέει εφόσον δεν μας δίνουν πληροφορίες οι εθνικές αρχές δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε χρονικά περιθώρια και προθεσμίες μέσα στις οποίες οι αρχές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να απαντούν. Διαφορετικά να υπάρχει ένας ε, μηχανισμός κυρώσεων. Φαίνεται ε, δυστυχώς πολύ αυστηρό κάτι τέτοιο, αλλά αν δεν υπάρχει αυτό το καθεστώς κυρώσεων, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη ανακύκλωσης. Τη στιγμή που στην Κίνα ανακυκλώνονται απόβλητα από την Ιαπωνία, που προέρχονται από την Ιαπωνία και μιλάμε για μια χώρα που έχει μεγάλα προβλήματα με τα απόβλητα, εμείς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αντιμετωπίζουμε επιφανειακά. Δηλαδή δεν υπάρχει βιωσιμότητα χωρίς ανακύκλωση των αποβλήτων. Δεν μιλάμε μόνο για πόντιση ή ρήψη αποβλήτων, αλλά θα πρέπει να ανακυκλώνονται σε χρήσιμα προϊόντα. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζονται αυστηρά κριτήρια και ουσιάδη, ουσιώδη κριτήρια με βάση τα οποία εμείς, τα κράτη-μέλη καθώς και οι περιφερειακοί φορείς να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Και άλλη μια φορά χαίρομαι για τη συνεισφορά όλων των συναδέλφων και της Τζούντιτ Μέρκης καθώς και των άλλων ομιλητών. Πιστεύω ότι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη νομοθεσία, διότι θα πρέπει με βάση τις οδηγίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας το πρόβλημά μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαβράκος. Ε, κυρία Πρόεδρε, η έκθεση είναι τόσο καλή που φοβάμαι ότι πρέπει να πάρουμε περαιτέρω μέτρα για να εφαρμοστεί. Διότι συνήθως τα καλά πράγματα δεν εφαρμόζονται και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τόσο <laughs> μεγάλο το θέμα και φύγει τόσο μεγάλα συμφέροντα και σε επίπεδο εταιριών αλλά και σε επίπεδο κακών κυβερνήσεων το λέω αυτό και γίνεται αντιληπτό τι λέω εις τρόπον ώστε μας επιβάλλει σε συνδυασμό με τις κοινωνικές αντιδράσεις που δημιουργεί όπου πάμε να φτιάξουμε έναν χιτά ή έναν ε, χώρο σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων. Μας επιβάλλει λοιπόν να βρούμε και συμπληρωματικά μέτρα ε, όπως θα ήταν η διεύρυνση της αρμοδιότητος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής, η χορήγηση ενός πιστοποιητικού ε, σε κάθε μελέτη από την Επιτροπή αυτή, εις τρόπον ώστε να ξεφύγουμε από τις νομικές διαδικασίες των ε, ε, δικαστηρίων των κατατόπους που δημιουργούν τεράστια προβλήματα χρόνου. Δηλαδή στην Ελλάδα που έχω μια εμπειρία, εάν προσφύγει κάποιος για έναν χιτά, θα έχει απόφαση μετά από πέντε χρόνια, δικαστική απόφαση μετά από πέντε χρόνια. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι στον ενδιάμεσο χρόνο πρέπει να γίνει μια διαχείριση των αποβλήτων και η διαχείριση αυτή να είναι και συνετή για το κοινωνικό σύνολο και ε, να είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης που ισχύουν σήμερα. Η ώστε να είναι ακίνδυνη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα και προς αυτίας μου επιτρέψει ο, ο κ. να του δώσω και ορισμένες σκέψεις μου στην, ε, μέχρι ότου έρθει στην Ολομέλεια τις οποίες ίσως θα συζητήσουμε και ίσως κάνει αποδεκτές για να δούμε πώς η ωραία αυτή η έκθεση θα γίνει αποτελεσματικότερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαίρω τον κύριο Ντουγκάζη για την καλή του έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος σε αυτήν την συζήτηση. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Σας υπενθυμίζω πάντως ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η τρίτη, η επόμενη τρίτη στις, στη μία το μεσημέρι ε, και φαντάζομαι ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις σας μπορούν ε, να μορφοποιηθούν σε τροπολογίες έτσι ώστε να βοηθήσουμε λίγο τον συνάδελφο ε, για αυτόν τον ε, βαρύ φόρτο που έχει με την έκθεσή του. έχουμε ήδη ε, ζητήσει και επίσης ε, να προχωρήσει κανονικά ε, η έκθεσή μας και σίγουρα στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Αν ο συνάδελφος Τουργκάης θέλει να πάρει το λόγο για κάποιες τελικές παρατηρήσεις, παρακαλώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις εξαιρετικές τους παρεμβάσεις, τις οποίες θα προσπαθήσω να εντάξω εδώ στην έκθεση. Θα αρχίσω από το τέλος, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Σαλαβράκος, δηλαδή σε σχέση με αυτές τις ιδέες ε, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν και όπως είπε και η Πρόεδρος γνωρίζουμε τις προθεσμίες μας. Ελπίζω αυτές οι ιδέες τις οποίες αναφέρατε να ενταχθούν σε τροπολογίες. Και χάρηκα πολύ για τον τρόπο που εκφραστήκατε. Μπορούμε να το συζητήσουμε εν είδη τροπολογιών Αλλιώς δεν, δεν μπορώ να πω ότι με, ενοχλεί να υποβάλλετε τροπολογίες. Είναι επικοδομητικές, αλλά ε, δεν θεωρώ καταρχήν ότι είναι ε, αρνητικό το να υποβάλλονται τροπολογίες. Και η Κομισιόν μίλησε για προβληματικά κράτη και γι' αυτό καταρτίζεται και αυτή η έκθεση. Αυτό θα ήθελα να πω και προς την ε, κυρία Μέρκης. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τους αναφέροντες αλλά και τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τους αναφέροντες που αναφέρουν τα συγκεκριμένα προβλήματα των κρατών. Όπως είπε και η Κομισιόν, πρόκειται για μία χαοτική κατάσταση. Δυστυχώς δεν συντάχθηκε πριν αυτή η έκθεση, θα μπορούσε να έχει συνταχθεί από εμάς, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όμως κάτι έπρεπε να γίνει για να καλυφθεί αυτό το κενό. Η κυρία Μέρκης μου είπε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τους αναφέροντες πρωτίστως και θα πρέπει να βρούμε ένα σχέδιο εφαρμογής. Δεν ξέρω ακριβώς τι ε, εννοούσατε, αλλά νομίζω ότι όταν μιλάμε για την έκθεση «Όκελ», για την αστιφιλία και τα προβλήματα του ε, τότε πρέπει κάπου να παραπέμψουμε τους πολίτες κάπου διότι ε, δεν υπάρχουν ε, πώς να το πω, προγράμματα πλαίσιο. Αυτό αφορά θέματα περιβάλλοντος, θέματα αστιφιλίας. Νομίζω λοιπόν ότι καλύπτουμε κενά και γι' αυτό χρειάζονται και αυτά τα σχέδια εφαρμογής. Εσείς ένα θέμα ουσίας ότι πολλές φορές δεν τηρείται και το γράμμα του νόμου. Και όταν δεν τηρείται το γράμμα του νόμου, συμβαίνει αυτό που βλέπουμε σε πολλά κράτη-μέλη, σε πολλές ε, κοινότητες. Δεν ξέρω ποιος το είπε. Νομίζω ότι ο κύριος Κωστινάρου, ο οποίος αποχώρησε, είπε ότι εάν δεν τηρείται ο νόμος, τότε θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, κίτρινες κάρτες, κόκκινες κάρτες, ό,τι θέλετε. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε το πλαίσιο κυρώσεων έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε και τους πολίτες και τα κράτη. Όπως έλεγε και ο Μιγκελάνχελ Μαρτίνες, εάν δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση ότι δεν πρέπει να μολύνουμε τότε δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι ο χρυσός κανόνας. Δηλαδή ότι καταρχήν δεν πρέπει να μολύνουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι ο χρυσός κανόνας και αυτό μπορεί να γίνει μέσω εκπαίδευσης. Θα ήθελα να τονίσω και το θέμα που έθιξε ο Αντιπρόεδρος, ο Μίγκελ Άγχελ. Ότι δηλαδή θα πρέπει το θέμα αυτό να το προωθήσουμε στην Ολομέλεια προς συζήτηση. Δεν θα πρέπει να το να υπεκφύγουμε αυτή της υποχρέωσης. Νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα και τις, μία από τις βασικές εκθέσεις της Επιτροπής μας και γι' αυτό θα πρέπει να τις προσδώσουμε τη, σημασία που της αρμόζει. Και νομίζω ότι ο Μίγκελ Άγχελ Μαρτίνες θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι απάντησα λίγο πολύ σε όλους έγινε λόγος και για υπέρβαση της νομοθεσίας και εδώ φέρουμε πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί πρόκειται για μία έκθεση μεγάλης εμβέλειας και ευθύνης για την Επιτροπή Αναφορών. Βεβαίω πρόκειται για επιμερισμένη ευθύνη. Δεν θα θέλαμε να εξατομικεύσουμε αυτή τη συζήτηση, απλώς να τη μετατρέψουμε σε μία ε, σοβαρή έκθεση, σε μία σημαντική έκθεση για τη σημασία που κατέχει. Είμαι στη διάθεσή σας και με μεγάλη μου χαρά θα δεχτώ όλες τις υποδείξεις και τροπολογίες που θα θελήσετε να μου υποβάλλετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συναδελφέ Τουργκάη. Ολοκληρώσαμε την εξέταση του σημείου αυτού. Περάμε στο επόμενο σημείο. Αναφυρά του κυρίου Αρκάντζελη, γαλλικής ηθαγένειας, για την διατήρηση της και την προστασία της ε, καφέ Αρκούδα στη Γαλλία. Είναι παρόν και θα του δώσουμε το λόγο για πέντε λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να ε, παρουσιάσω αυτήν την ε, έκθεση, την αναφορά, συγγνώμη, η οποία ε, αποτελεί κοινή αναφορά 15 γαλλικών ενώσεων για την προστασία της Αρκούδας. Λέγομαι Φρανσουά Αρκαντζελή, είμαι πρόεδρος της οργάνωσης Paydours η δήμαρχος της Αρμπάσα στην Οτ Γκαρόν και περιφερειακό σύμβουλο στα Μιντή Πυρενέ στην Νοτιοανατολική Ανατολική ε, Γαλλία ε, στην, ε, στα, στους αριθμούς 92-43 της οδηγίας οικότοπη Habitat αναφέρεται το είδος το υποδιατήρηση της καφέ αρκούδας Ούρσους Άρκτος. Ε, και βεβαίως ε, σκοπός και στόχος είναι να διατηρηθεί ο οικότοπος ε, της καφέ Αρκούδας καθώς επίσης και ικανός πληθυσμός. Στη, στα Πυρηναία ο πληθυσμός των καφέ Αρκούδων βρίσκεται στις δύο πλευρές του και σε δύο υποπληθυσμούς. Τον δυτικό υποπληθυσμό που έχει μονάχα δύο αρσενικές αρκούδες και στο, σε αυτόν τον τομέα των Πυρηναίων που μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ εξάλληψη του είδους. Ε, δυστυχώς τα μέτρα ήταν πολύ δειλά και ε, οπωσδήποτε δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να βρίσκεται σχεδόν υπό εξαφάνιση. Επομένως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναπλαστεί ο πληθυσμός σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει επίσης ο πληθυσμός στα κεντρικά και ανατολικά Πυρηναία που είχαν ελευθερωθεί αρκούδες το 1996-1997 και το 2006 ε, και υπάρχουν και οι απόγονοί τους. Το 2010 είχαμε 16 ε, αρκούδες, 3 αρσενικές, 5 ε, θηλυκές σε όριμη ηλικία καθώς και 2 πριν την ηλικίωση, 4 μικρά αρκουδάκια καθώς και 2 ακαθόριστα ήδη. Ε, αυξάνεται ο πληθυσμός κατά μία αρκούδα ανά έτος. Ε, μονάχα μία αρκούδα πέρασε, αρσενική μάλιστα, πέρασε από τη μία περιφέρεια στην άλλη στα 15 τελευταία χρόνια. Αυτοί οι δύο υποπληθυσμοί είναι επομένως ε, ε, ε, ξεχωρισμένοι και η Εθνική Υπηρεσία Κυνηγιού και Άγριων Ζώων πάντα τις μελετούσε ξεχωριστά. Το 2005 η μελέτη βιωσιμότητας της αρχής την οποία ανέφερα προηγουμένως είχε καθορίσει ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν τουλάχιστον 9 αρκούδες στα δυτικά Πυρηναία και τουλάχιστον 4 ε, στα ε, κέντρο ανατολικά έτσι ώστε να είναι βιώσιμο το είδος. Όμως ε, μονάχα 5 αρκούδες από τις 13 που ήταν απαραίτητες τελικά απελευθερώθηκαν το 2006 και μονάχα στα κεντρικά Πυρηναία μονάχα 4 ήταν φιλικές, 2 πέθαναν πρώιμα ε, και η μία δεν απέκτησε ποτέ απογόνους. Ε, σύμφωνα με την μελέτη του 2009, δηλαδή μετά και τις απελευθερώσεις του 2006, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε για να είναι βιώσιμος ο πληθυσμός να απελευθερωθούν ακόμα περισσότερες αρκούδες, 16 στα δυτικά Πυρηναία και 4 στα κέντρο-ανατολικά Πυρηναία. Ε, και σύμφωνα με την τελική μελέτη του 2009 βρίσκεται ο πληθυσμός σε κρίσιμο σημείο κινδύνου εξαφάνισης. Το 2011 καμία, κανένας από τους δύο υποπληθυσμούς δεν ήταν σε καλό σημείο διατήρησης. Ε, όσον η ε, γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε παρόλα αυτά να μην, ε, να μην απελευθερώσει άλλες αρκούδες και απλώς να έχει μια στρατηγική προστασία της βιοπικιλότητας. Όσον αφορά τις καφέ αρκούδας δεν έχουμε στοιχεία που να μας οδηγούν ότι πραγματικά θα υπάρξει αποκατάσταση των πληθυσμών. Ε, αντιθέτως ε, η κυβέρνηση μετά από την πίεση του λόμπι των ε, γεωργών αποφάσισε να μην, να μην προχωρήσει στην διατήρηση του, της αυτού του πληθυσμού των αρκούδων. Η κατάσταση της καφέ Αρκούδας ε, στην ε, Γαλλία είναι σε κρίσιμο σημείο πλέον, ιδιαίτερα στα δυτικά Πυρηναία και η Γαλλία δεν έχει πλέον καμία πολιτική διατήρηση του είδους εδώ και ε, πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από το 2009. Η Γαλλία επίσης δεν σέβεται την οδηγία 92 92-43, την λεγόμενη οδηγία οικοτόπων, κυρίως δε το άρθρο 12 και επίσης και το άρθρο 22 όπου αναφέρονται τα κράτη-μέλη μελετούν την σκοπιμότητα Απελευθέρωση ειδών του, του παραρτήματος 4 αυτόχθονα ε, στο, στην περιφέρεια ε, εάν το μέτρο αυτό μπορεί να συμβάλλει στην συντήρησή τους. Πολλές ε, αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κατατεθεί από τις, από τις υπηρεσίες αρμόδιας καθώς επίσης και από τις διάφορες ε, ενώσεις ε, και συγκεκριμένα το 2009 είχαν ε, υποβληθεί δύο αναφορές οι οποίες όμως έμειναν χωρίς καμία, καμία συνέχεια. Επίσης σε απάντηση σε ερώτηση που προσφάτως έθεσε η κυρία Σαντρίν Μπελιέ στην Επιτροπή όσον αφορά την στρατηγική των πυρηναίων και την βιοπικιλότητα πρέπει να πούμε ότι και αυτή η ερώτηση παρέμεινε ανα απάντητη. Βεβαίω, όσον αφορά το θέμα τη ε, βιοπικιλότητα, ε, μαζί θα πρέπει να δούμε και την οικονομική ανάπτυξη αυτών των ορεινών περιοχών. Ε, και βεβαίω, πέρα από την μείωση τη της ποικιλία των ειδών, η εξαφάνιση του, ε, του είδους της ε, καφέ αρκούδας ε, μπορεί να σημάνει και μείωση των τουριστών καθώς επίσης και μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και οπότε των εισόδων αυτών των περιοχών που ήδη αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αρκάντζελη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε δύο εκπροσώπους. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Γκριμού. Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι αναφέροντες, καλημέρα σας. Ε, χαίρομαι που έχουμε σήμερα την ε, δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα το, της καφέ Αρκούδας στα Πυρηναία. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η αναφορά αυτή ε, ε, πραγματικά φέρνει το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οροσυρά ε, αλλά πρόκειται και για ένα είδος το οποίο κατά προτεραιότητα απασχολεί τους Ευρωπαίους πολίτες, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα όμως τώρα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο από την ε, ε, ε, διεύθυνση της φύσης Nature και ο οποίος θα αναφερθεί στα μέτρα τα οποία έχουν αναλυφθεί, τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί τα τελευταία χρόνια από τις γαλλικές αρχές όσον αφορά την οροσυρά των πυρηναίων έτσι ώστε να διατηρηθεί η βιοπικιλότητα και έτσι ώστε και η καφέ αρκούδα να παραμείνει βιώσιμο είδος είναι γεγονός ότι η Γαλλία ε, αποφάσισε να μην απελευθερώσει ε, μία θηλυκιά αρκούδα στα δυτικά Πυρηναία ε, και πραγματικά πήρε τελευταία κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα αναφερθούν στην έποψη αυτή, την επισκόπηση μάλλον των μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως όχι μονάχα ενδιαφέρεται για το θέμα ε, στα πλαίσια αυτής της αναφοράς αλλά και βάσει οκτώ ε, μηνύσεων που έχουν υποβληθεί για το θέμα ε, αυτό και οι οποίες επισήμως έχουν καταγραφεί ε, εις το σύστημα CHAP που είναι το σύστημα καταγραφής ε, των ε, προσφυγών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί και στην ετήσια συνάντηση που έχουμε με τις γαλλικές αρχές στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουμε για τις προσφυγές και για τα σημεία τριβής. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι με μεγάλη προσοχή μας απασχολεί το θέμα αυτό. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμόσει οι γαλλικές αρχές τα τελευταία χρόνια. Πρώτα απ' όλα και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως υπήρξε μια προσπάθεια εν πάση περιπτώσει των γαλλικών αρχών ε, να ανακόψουν την ε, ε, μειωτική πορεία του πληθυσμού της καφέ Αρκούδας. Το 1995 δεν υπήρχε καμία αρκούδα ε, το κέντρο ανατολικό πυρήνα ε, και ε, πολύ λίγα και πολύ λίγα ζώα στον κέντρο δυτικό πυρήνα. Το 1996-97 και το 2006 απελευθερώθηκαν αρκούδες στο κεντρικό και ανατολικό πυρήνα Οχτώ συγκεκριμένε αρκούδες ε, απελευθερώθηκαν οι οποίε προέρχονται από την Σλοβενία στα πλαίσια μιας διμερούς ε, συμφωνίας ε, μεταξύ των δύο χωρών. Οκτώ λοιπόν αρκούδες απελευθερώθηκαν σε έναν από τους ε, πυρήνες ε, και ο οποίος σήμερα αποτελείται από 17 έως 19 ε, ζώα μεταξύ των οποίων και θηλυκές οι οποίες γέννησαν νεογνά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το πρώτο έτος της ηλικίας τους και επομένως θεωρούνται βιώσιμα. Ε, στον άλλο πυρήνα, ο οποίος είναι και πιο ε, προβληματικός, εκεί έχουν παραμείνει μονάχα αρσενικά ζώα. Αυτό σημαίνει ότι ελήψη θηλυκών δεν θα υπάρχει αναπαραγωγή και επομένως ε, κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ζώα, χωρίς αρκούδες καφές αυτόν των πυρήνα. Οι αναφέροντες αναφέρθηκαν στο άρθρο 12 συγκεκριμένα. Πρέπει να πούμε λοιπόν επ' αυτού ότι οι γαλλικές αρχές έχουν ε, εκπονήσει ένα πρόγραμμα διατήρησης ε, των, της καφέ Αρκούδας 2006-2009. Ένας τρόπος προστασίας των, της Αρκούδας είναι η προστασία του οικότοπου ε, της Αρκούδας. αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει καθορίσει πέντε ε, περιφέρειες ε, Natura 2000 ε, που αποτελούν οικότοπο της Αρκούδας. Άρα εφαρμογή του 6234 έχει ήδη αρχίσει να ισχύει το νομικό καθεστώς προστασίας των οικοτόπων. Επίσης οι αναφέροντες έχουν ε, αναφερθεί σε ένα άρθρο το οποίο ε, πλέον δεν εφαρμόζεται. Ε, συγγνώμη, αναφέρθηκαν σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης της βιοπικιλότητας το οποίο πλέον δεν ισχύει. Οι γαλλικές αρχές τις οποίες στράφημεν όντως μας είπαν ότι δεν ε, ε, εφαρμόζεται το άρθρο αυτό ε, και ότι προτίθεντο να απελευθερώσουν μια θηλυκιά αρκούδα έτσι ώστε να υπάρξει εκ νέου αναπαραγωγή στον πυρήνα που δεν είχε θηλυκιά για την ώρα, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και περιμένουμε από τις γαλλικές αρχές να μας ενημερώσουν για το θέμα αυτό. Ε, επίσης υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην καφέ Αρκούδα και τις συμφωνίες ε, κυνηγιού. Ε, στην συγκεκριμένη περιφέρεια καθορίζεται νομοθετικά ότι τρόπος και η αντιμετώπιση της, της, ε, του κυνηγιού σε περιοχές ε, παρουσίας ε, της καφέ αρκούδας. Σύμφωνα με τα, με επαρχιακά διατάγματα λοιπόν και σε, σε περίπτωση ανείχνευσης παρουσίας καφέ αρκούδας σταματάει το κυνήγι στην περιοχή αυτή. Ε, επίσης υπάρχουν ε, και κάποιες ε, συμφωνίες όσον αφορά την παρουσία της καφέ αρκούδας και τη γεωργία συγκεκριμένα δε τα βοσκοτόπια. Ε, τις ε, τελευταίες, ε, τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προστασίας των κοπαδιών, των κτηνοτρόφων από τις καφέ αρκούδες. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια απόκτησης ειδικών τσοπανόσκυλων κτλ. Όπως σα έλεγα προηγουμένως, πολλές προσπάθειες καλής διαχείρισης της κατάστασης ε, έχουν εκπονηθεί ε, και βεβαίω θα δώσω αμέσως το λόγο στον συνάδελφο Μάρκο Τσιπριάνη, ο οποίος ε, θα μας πει ακριβώς περί τίνο πρόκειται. Ευχαριστώ να κάνω και εγώ κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά την κατάσταση διατήρησης. Το να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο διατήρησης για όλα τα ήδη αποτελεί τον απότερο στόχο της οδηγίας αυτής. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η οδηγία δεν θέτει προθεσμία για τους στόχους αυτούς και η οδηγία ορίζει ότι τα μέτρα για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Αυτά θα καθορίσουν το πώς θα το πετύχουν, πώς θα πετύχουν τα αποτελέσματα αυτά. Και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οι οικονομικές και ε, πολιτισμικές πτυχές, αλλά και τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά. Αυτά ορίζονται στο άρθρο 2. Τώρα, το... η κατάσταση διατήρησης θα πρέπει να αξιολογείται βάσει τριών παραγόντων. Η δυναμική του πληθυσμού, ε, η φυσική ποσόστοση και ο οικότοπος. Η δυναμική του πληθυσμού υποδεικνύει ότι είναι βιώσιμος πυρήνας ε, που μπορεί από μόνος του να συντηρηθεί στον ε, βιότοπό του. Άρα δεν θα μειωθεί κατά πάσα πιθανότητα ε, το ποσοστό του είδους τα επόμενα χρόνια. Και τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές, ένας επαρκής βιότοπος σε έκταση για να φιλοξενεί το είδος. Αυτό είναι ο ορισμός ε, της ε, οδηγίας. Στις σχετικές οδηγίες που έχουμε εκδώσει, έχουμε δώσει περισσότερα στοιχεία, περισσότερες λεπτομέρειες για τα μεγάλα σαρκοφάγα ζωά και να δούμε τι έχει γίνει για την αξιολόγηση αυτού, αυτής της κατάστασης διατήρησης του είδους. Στο άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους ορίζονται τα σχετικά κριτήρια. έγινε μια πρώτη αξιολόγηση των ειδών και των βιοτόπων από την οδηγία. Τώρα, η εκτίμηση για τις αρκούδες στα γαλλικά πυρηναία. Βλέπουμε από την έκθεση που λάβαμε από τις γαλλικές αρχές ότι εκτιμάται ότι ο πληθυσμός, η δυναμική του πληθυσμού και οι μελλοντικές φρουτικές είναι μάλλον μη ευνοϊκές. Κάποια συμπεράσματα λοιπόν από πλευρά μα. Τι συμπεράσματα μπορούμε να εξαγάγουμε. Καταρχά, σαφώ βελτιώθηκε η κατάσταση από τότε που εφαρμόστηκε ε, η οδηγία για τους οικοτόπους. Να λάβουμε υπόψη ότι το 94, από το 94 μάλλον, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί από 5 άτομα σε 20 άτομα, σε 20 αρκούδες και αυτό οφείλεται σε δύο μέτρα, το 96 και χάρη σε μέτρα που προωθούν και ενθαρρύνουν την ε, συνύπαρξη την, με τις ανθρώπινες ε, δραστηριότητες για τη διατηρήση των αρκούδων. Άρα, υπήρξε βελτίωση από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία. Κατά δεύτερον, διαπιστώνουμε ότι δεν αρκούν αυτές οι προσπάθειες που έγιναν, γιατί η κατάσταση της διατήρησης δεν είναι επαρκής. Άρα χρειάζεται παραπάνω προσπάθεια. Ξέρουμε λοιπόν, μέχρι το 2009 είχαμε το σχέδιο για την ανοικοδόμηση του, για την ανασύσταση του πληθυσμού. Ε, από τότε και μετά δεν ξέρω να υπάρχουν νέα τέτοια σχέδια, αλλά θα διαβουλευτούμε και με τι γαλλικέ αρχέ. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Δεν ξέρω, ένας ομιλητής έχει ζητήσει το λόγο. Μία ομιλήτρια μάλλον, η οποία έχει το λόγο και είναι και η τελευταία στον κατάλογο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να επανέλθω στη συζήτηση, αλλά με εκπλήσει η παρέμβαση της Επιτροπής. Γιατί μιλάμε για παραβίαση της οδηγίας για τα οικοσυστήματα. Το κείμενο είναι απόλυτα σαφές, το κείμενο της οδηγίας. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να ορίσουν ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας των υποεξαφάνιση ειδών, δηλαδή στην περίπτωση αυτή της καφέ αρκούδας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κατάσταση μέσα στα πλαίσια της συντήρησης αυτού του είδους. Σήμερα το γαλλικό κράτος, το λένε και αναφέρονται στο λέει και Κομισιόν. Από το τέλος του 2009 η Γαλλία δεν διαθέτει σχέδιο συντήρησης ή αποκατάστασης των πυρηναίων, υπάρχει νομικό κενό, άρα δεν έχουμε κανένα σύστημα προστασίας εδώ και δύο χρόνια, όπως ορίζει η οδηγία για τα οικοσυστήματα. Άρα από το 2009 η Γαλλία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις, άρα παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Για το δεύτερο σημείο η Επιτροπή μας λέει ότι από το 1992-1994 υπάρχει μία μικρή βελτίωση. Δηλαδή η κατάσταση των αρκούδων είναι λίγο καλύτερη. Αλλά δεν μιλάμε για λίγο καλύτερη κατάσταση και μόνο τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση, έχουν υποχρεώσεις αποτελεσμάτων. Δεν μιλάμε για βελτίωση της κατάστασης, αλλά για μια κατάσταση συντήρησης και αποκατάστασης για ένα είδος το οποίο βρίσκεται υπό εξαφάνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα μας λέει η Επιτροπή ότι η Γαλλία δεν μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο για τα Πυρηναία. Υπ' αυτές τις συνθήκες και επειδή δεν υπάρχει αυτός ο πυρήνας σύντηρησης, δεν θα σας πω εγώ πώς ε, λειτουργεί η φύση και πώς πρέπει να συντηρήσουμε έναν πληθυσμό, ζωικό πληθυσμό. Δεν θα αρχίσουμε με μάθημα, με ένα μάθημα βιολογίας, αλλά θα ήθελα να πω ότι η οδηγία αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα συντήρησης έτσι ώστε να μην θανατώνονται και να μην φυλακίζονται τα ίδια αυτά. Από το 2005, εδώ και έξι χρόνια, βλέπουμε ότι θανατώθηκε και το τελευταίο θύλι Άρα, εδώ και πέντε χρόνια δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο και γι' αυτό θα πρέπει να εισαγάγει ένα θύλι την Άνοιξη του 2011. Και αυτό είναι το ερώτημά μου προς την Κομισιόν. Πώς έχει η κατάσταση ε, γιατί οι δεσμεύσει της Γαλλίας δεν ή μάλλον η Γαλλία δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της. Άρα η βιωσιμότητα της καφέ αρκούδας δυναμητίζεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε αμφίσιμες απαντήσεις. Τον Ιούλιο του 2011 διαμέσου του Επιτρόπου Ποτότσνικ οι απαντήσεις ήταν λίγο πιο σαφείς. Θα ήθελα να δείτε τις απαντήσεις του Επιτρόπου Περιβάλλοντος για την κατάσταση στη, της Γαλλίας, διότι η Γαλλία παραβιάζει το δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο ως προς την κατάσταση της αρκούδας των Πυρηναίων, άρα δεν μπορεί να διευθετηθεί η κατάσταση και δεν υπάρχουν εγγύησεις. Τι πρέπει να γίνει σήμερα. Πόσο καιρό, πόσος καιρός πρέπει να περάσει κατά την Κομισιόν. Γιατί η οδηγία για τα ενδιαιτήματα προβλέπει ανά έξι χρόνια ε, εξέταση. Δηλαδή 98, 2004, 2010. Σήμερα έχουμε εγγυήσεις για τη βιωσιμότητα της κατάστασης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, χρειάζονται περαιτέρω αξιολογήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει η συντηρητική αρχή της βιοπικιλότητας έτσι ώστε οι γαλλικές αρχές να πρέπει να οφείλουν να αντιδράσουν. Και θα ήθελα στην Επιτροπή μας να ξαναθίξουμε αυτό το θέμα στο τέλος του 2011 για να δούμε κατά πόσο η Γαλλία θα έχει ανταποκριθεί μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα κρατάμε ανοιχτή αυτή την ε, αναφορά μέχρι το τέλος του έτους. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν το λόγο, κάποιος άλλος. θα δώσουμε το λόγο για άλλη μία φορά στους αναφέροντες έτσι ώστε να απαντήσουν με βάση αυτά που άκουσαν, αν το επιθυμούν. Όπως θέλετε. Αν θέλετε μπορείτε να λάβετε το λόγο. Όχι. Ενδεχομένως ε, θα μπορούσα να επιμείνω λίγο περισσότερο αλλά είναι γεγονός ε, ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες ε, ε, συμπίπτουν στην ίδια διαπίστωση ότι δηλαδή δεν υπάρχει σωστή διατήρηση του πληθυσμού και μάλιστα θα πρέπει να απελευθερωθούν 17 δείγματα του είδους έτσι ώστε να έχουμε ελπίδα διατήρησης του ε, πληθυσμού. Εμείς από την πλευρά μας απλώς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αναφέροντα έχοντας ακούσει όλα ε, τα ζητήματα να ε, φαντάζομαι να συμφωνείτε ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες από την γαλλική ε, από το γαλλικό κράτος έτσι ώστε να έχουμε περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως είναι το σημείο 9 Πρόκειται για αναφορά της κυρίας Λάουρα Di Καρλ Αντώνιο, Ιταλικής Ιθαγένειας, σχετικά με απαγόρευση κυνηγιού της καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία. Παρακαλώ. Η κυρία Σίλβια Βαραβά θα ε, πάρει το λόγο ξενόδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Bonjour. Ναι, θα αντικαταστήσω εγώ τον συνάδελφό μου. Κανένα πρόβλημα. Ο αναφέρον ζητά να γίνει επαγόρευση της, ε, του κυνηγιού της Αρκούδας στη Βουλγαρία. Υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα προστατευμένο είδος, όπως είπαμε και για το προηγούμενο σημείο της ημερήσιας Όντως πρόκειται για ένα είδος υποπροστασίας, ε, αλλά η οδηγία ορίζει διάφορες εξαιρέσεις τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κρατη σε περίπτωση που θέλουν ε, να επιτρέψουν το κυνήγι κάποιων ατόμων του είδους. Και αυτό συνέβη στη Βουλγαρία. Λάβαμε λοιπόν τη σχετική καταγγελία. Ξεκίνησε έρευνα προσκειμένου να τεθούν ερωτήσεις στις βουλγαρικές αρχές για να δούμε κατά πόσον πληρούνται όλες οι, όλοι οι όροι για τις εξαιρέσει ε, που ορίζει η οδηγία. Ε, στην παρούσα φάση αναμένουμε ακόμα απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος ζήτησε το λόγο. Φαίνεται ότι εμπειρογνώμονες, είσαστε εμπειρογνώμων για θέματα αρκούδας. Mm. Όχι. Θα πρότεινα μόνο οι Βούλγαροι εάν θέλουν να, μην έχουν πια αρκούδες να τις στείλουν στη Γαλλία. Έτσι θα έχουμε δύο αναφορές στην τιμή της μίας. Θα είχαμε μία συνεργασία Βουλγαρίας-Γαλλίας. Προτείνω να ε, παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά εκκρεμούσα δηλαδή μέχρι ότου μας ενημερώσει η Βουλγαρία. Αλλά ως προς συνεργασία Βουλγαρίας-Γαλλίας νομίζω ότι ίσως θα μπορούσαμε έτσι να λύσουμε και τα δύο θέματα. Υπάρχει κανείς που ζητάει το λόγο. Δεχόμαστε με την υπόδειξη της κυρίας Μπελιέ. Την υπόδειξη της κυρίας Μπελιέ περνάμε στο 10 αναφορά του Μανουέλ Αντώνιο Καουπράδο, Ισπανικής Ιθαγένης, εξ ονόματος συντεχνίας αλλιέων της ε, Κορούνια, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές ενώσεων. Για την μόλυνση της περιοχής Ρίαντεμπουργού. Καλό σας απόγευμα, σας δίνω το λόγο. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ που μας λάβετε υπόψη. Εκπροσωπούμε την περιοχή της Κορούνια. Ερχόμαστε από τη Γαλλικία για να σας αναπτύξουμε αυτό το θέμα που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Μετά από πολλές καταγγελίες και διαμαρτυρίες και εδώ και στις Βρυξέλλες ξεκίνησαν προσφυγές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσάς και ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπόψη την αναφορά μας επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα θέμα μόλυνσης των υδάτων και ιδιαίτερα ευρωπαϊκών υδάτων. Πώς έχουν τα πράγματα. Η Ντεβούργο, όπως ξέρετε είναι μία ε, περιοχή μεγάλης παραγωγής, παραγωγής και ε, αλίας. Και δυστυχώς στη δεκαετία του 90 περάσαμε από 2.167 αλίες σε μόνο 130 αλίες. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και 20 χρόνια η κατάσταση ρήψη των αποβλήτων έχει οδηγήσει εδώ και 20 χρόνια σε μεγάλες επιπτώσεις στην, ε, ε, στις θέσεις εργασίας, δηλαδή στην απασχόληση, αλλά και στις ποιότητες των υδάτων, διότι υπάρχει μεγάλη μόλυνση της οικονομικής και παραγωγικής αυτής ζώνης, δηλαδή της παράκτιας αυτής γραμμής. Παρά τις ε, καταγγελίες που έχουν γίνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, δυστυχώς οι τοπικές αρχές δεν έχουν επιβάλει κανένα μέτρο. Το 1996 η κοινότητα της Γαλλικίας μίλησε για την εξυγίανση της περιοχής και τη βυθοκόρηση της περιοχής, μιλώντας για 78 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδότηση από την Ευρώπη. Ως προς τα ε, απόβλητα, τα αστικά απόβλητα, δυστυχώς ποντίζονται στις εκβολές του ποταμού του Μπούργου, χωρίς να γίνεται καθαρισμός των υδάτων και χωρίς να υπάρχει εγκατάσταση καθαρισμού. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, δυστυχώς η πόλη της ε, Κορούνια δεν είναι η μόνη πόλη που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Έχει 200.000 ε, κατοίκους και μέχρι σήμερα δεν έχει καμία εγκατάσταση καθαρισμού για τα υπολοιματικά ύδατα και δυστυχώς και οι όμορες περιοχές με 100.000 κατοίκους αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα. Η δυσμενής αυτή κατάσταση σχετίζεται και με την υγειονομική ταφή βιομηχανικών προϊόντων σε σχέση δηλαδή με σφάγια τα οποία ρίπτονται, φυτοφάρμακα και υπολείμματα σαπουνιών και δυστυχώς δεν υπάρχει και αποχετευτικό δίκτυο το οποίο να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση ολιστικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια αντιμετώπισης χώρων υγειονομικής ταφής. Επειδή έχουν γίνει πολλές προσφυγές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος του Δήμου της Γαλλικίας και επειδή δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια εξυγίανσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη επιπροσθέτως το γεγονός ότι εδώ και έξι μέρες έγινε πόντιση 35.000 λίτρων κυροζίνης στις εκβολές του Μπούργο και εδώ και πέντε μέρες ε, μία άλλη πόντιση 70.000 λίτρων αποβλήτων υπονόμων από τον Δήμο του Κουγερέδο. Άρα έχουμε ένα υψηλό επίπεδο μόλυνσης των υδάτων. Αυτό διακυβεύει την υγεία των πολιτών καθώς και τη μόλυνση των εκβολών του Μπούργο. Εάν δεν επιληθεί αυτό το πρόβλημα δεν βλέπουμε μέλλον. Γι' αυτό ζητούμε να εφαρμοστούν τα κατάλληλα νομικό μέτρα, νομικά μέτρα και να προβλεφθεί ένα συνολικό πρόγραμμα εξυγίανσης της περιοχής της Ρία. Δηλαδή ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά μέχρι ότου ε, προβλεφθεί κάποιο είδος επίλυσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεταβεί στη Γαλλικία για να δει πώς έχει κατάσταση στην περιοχή της Ρίαντελμπουργκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους αναφέροντες και την ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ε, μιλώ εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, γιατί θεωρούμε ότι η νομοθεσία για την προστασία των υδάτων έχει μεγάλη σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και για τον υδροφόρο ορίζοντα. Υπάρχει ένας, ε, υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις δυνάμει της οδηγίας για τα ύδατα και θεωρούμε ότι μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχει γίνει σχετικός τουλάχιστον καθαρισμός υδάτων. Πιστεύω ότι ο κοινός παρονομαστής μας θα πρέπει να είναι ο καθαρισμός υδάτων σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε κρατικό έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στην ανάλυση των προβλημάτων καθώς και να προβάλλουμε μέτρα επίλυσης. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε τα μέτρα για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για τα υπολοιματικά αστικά ύδατα. Χωρίς αυτά τα μέτρα, από τεχνικής πλευράς, είναι αδύνατον να υποβοηθήσουμε το περιβάλλον θα πρέπει να μιλήσουμε για βασικές ζώνες όπου υπάρχουν παραγωγικές δραστηριότητες όπως η αλία σε επίπεδο παράκτιων περιοχών. Και θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έλαβε μέτρα κατά του Ισπανικού κράτους που ε, ε, δεν πληρεί αυτούς τους τρεις όρους που σας προανέφερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προσφυγή στο ΔΕΚ κατά της ε, Ισπανίας για τα μέτρα που δεν έλαβε, δηλαδή για τον καθαρισμό των θαλασσών. Και με βάση αυτή τη διαδικασία, ήδη τον Ιούλιο έγινε η προσφυγή κατά της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μετά από καταγγελία λοιπόν της Κομισιόν το 10 καταδίκασε την Ισπανία για παραβίαση της νομοθεσίας περί πολυματικών υδάτων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου διαπιστώσαμε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις η Ισπανία και στην περίπτωση της Κορούνια έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο αστικό κέντρο με ένα πληθυσμό άνω των 250.000 όπου δεν υπάρχει σωστή διαχείριση των υπολοιματικών υδάτων. στα πρώτα βήματα αυτής της αναφοράς που έχει μεγάλη ιστορία, έχει προϊστορία εδώ, Θεωρήσαμε ότι η περιφερειακή κυβέρνηση θα πρέπει να προβάλλει ένα σχέδιο βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων όπου υπάρχει παραγωγή ε, μαλακοστράκων. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβληθούν συγκεκριμένα μέτρα μετά από απόφαση του ΔΕΚ και ελπίζουμε ότι αργά ή γρήγορα το ΔΕΚ θα καταδικάσει την Ισπανία και στη νέα μας αυτή προσφυγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιτουργκάης έχει το λόγο. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να καλωσορίσω και εγώ τον ε, συμπατριώτη μου. Όπως ξέρετε, πρόκειται για μία περιφέρεια στην οποία προσδώσαμε μεγάλη σημασία και καταβάλαμε πολλές προσπάθειες βελτίωσης, αλλά όπως ξέρετε είχαμε και μια περιβαλλοντική καταστροφή, δηλαδή ένα φορτηγό έριξε το φορτίο του στις εκβολές αυτές και βλέπουμε ότι πολλές φορές πλήττεται το περιβάλλον και το είδαμε για άλλη μια φορά στις εκβολές. Θα ήθελα κάθε οργανισμός να ανταποκρίνεται στο, στο έργο του και αυτό αφορά και τις τοπικές αρχές. Θα ήθελα να σας πω ότι από πλευρά της κοινότητας της Γαλλικίας στις εκβολές αυτές και στη ζώνη αντιμετωπίσαμε προβλήματα γιατί μιλήσαμε για εξυγίαση του Μπούργου, για καλύτερη ε, αντιμετώπιση των ε, υπολοιματικών υδάτων, για αντιμετώπιση των αναχωμάτων και των αμολόφων και ούτω καθεξής. Έγινε λόγος για 10 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό στην περιοχή των εκβολών του Μπουργό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη μόλυνση αν και βλέπουμε ότι οι επενδύσεις έχουν αυξήθει. Αλλά όλα εξαρτώνται από την καλή ε, διαχείριση των τοπικών αρχών και των προγραμμάτων εξυγίανσης. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν και οι μελλοντικές επενδύσεις θα αντιμετωπίσουν και το θέμα των υγειονομικών ταφών έτσι ώστε να μην γίνεται πόντιση στις εκβολές. Ο κύριος Θαπατέρο, οι κύριοι Θαπατέρο και Μπλάνκο θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα των βιομηχανικών μονάδων που βρίσκονται πολύ κοντά στην παράκτια περιοχή. Αυτό μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Υπήρχαν παρόμοιες αναφορές και στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους υπήρξε ένα κονδύλι το οποίο όμως ε, δεν εκτελέστηκε. Δεν εκτελέστηκε δηλαδή ο γενικός ε, προϋπολογισμός. Και δυστυχώς εξαφανίστηκε και από τον προγραμματισμό υπάρχει και μία διαδικασία που εκρεμεί ενώπιον ε, του ΔΕΚ. Πρόκειται για προσφυγή της Κομισιόν. Και όπως είπα και πριν, θα πρέπει να δούμε τι, κάνει, τι κάνουν οι δημοτικές αρχές για την εξυγίανση των εκβολών και τις παράκτιες ζώνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η κατάσταση που μόλις μας ε, εξετέθη είναι ε, απαράδεκτη, δεν μπορεί κανείς να τη φανταστεί. Είναι πέραν κάθε φανταστίας ε, για μια ευρωπαϊκή χώρα. Κυρίως όταν ε, υπάρχουν παλαιές νομοθεσίες όσον αφορά την προστασία των υδάτων. Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν επί ευρωπαϊκού εδάφους να εξακολουθούν οι υφίστανται τέτοιες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στο ότι υπάρχει ε, καταδίκη της Ισπανίας στις 14 Απριλίου του 2011 ε, και ότι επομένως η χώρα αυτή θα υποχρεωθεί να υποβάλει ε, και να επιβάλλει τα απαραίτητα μέτρα. Επομένως, συμφωνώ να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, αλλά ενδεχομένως να πάμε παραπέρα, να ζητήσουμε και επιτόπου αποστολή της ε, Επιτροπής μας ε, έτσι ώστε να δούμε λίγους μήνες μετά με ποιο τρόπο ε, προσπαθεί να ε, αντιμετωπίσει η Ισπανία μια καταδίκη την οποία δέχθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Α, υπάρχει μήπως θέλει ο αναφέρον να ξαναπάρει το λόγο. Ε, κύριε Καου, Καουπράδο, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πράγματι είναι σουρεαλιστικό το σενάριο, όπως είπε η κυρία πελίε. Εγώ ζω αυτή την κατάσταση καθημερινά θα ήθελα να το ξέρετε, σας δείχνω πώς έχει η κατάσταση στις εκβολές του Μπούργο με όλα τα σημεία ρήψεων. Πρόκειται για μία εκβολή ε, μεγάλης ε, εμβέλειας, το 25% το, της αλίας γίνεται εκεί και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επειδή πρόκειται για μια τόσο μεγάλη έκταση, η κατάσταση επιδεινώνεται. Εδώ σας δείχνω μια άλλη φωτογραφία. Όταν ήμασταν 2.160 αλείς, σήμερα είμαστε μόνο 130. Έχουμε μια συντεχνία, πρόκειται για πολλούς νέους που θα ήθελαν ένα μέλλον. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπωσδήποτε κατά αυτήν την έννοια και προς, ε, προς την βοήθεια την οποία ζητάτε ε, οδεύουν ακριβώς ε, και οι παρεμβάσεις των συναδέλφων. Παραμένει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά. Πρέπει να σας πω ότι έχω και μια ανακοίνωση από, την, από τον που ακριβώς υπογράμμιζε το ενδιαφέρον το οποίο κατά την άποψή του ε, έχει αυτή η αναφορά την οποία ε, ζητά και να παραμείνει ανοιχτή μέχρι ότου να ολοκληρωθούν ε, και οι δικαστικές διαδικασίες καθώς επίσης και να ολοκληρωθεί και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα, την πρόταση της κυρίας Μεριά οπωσδήποτε σχετικά με επιτόπου αποστολή σε, στην επόμενη συνεδρίαση των ε, συντονιστών μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ε, δεν ξέρω εάν φέτος θα βρούμε χρόνο, αλλά πάντως μπορούμε το 2012 να εγγράψουμε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίσκεψης επιτόπου. Ε, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αναφέροντα. Περνάμε στην επόμενη αναφορά. Είναι η αναφορά του, που έχει υποβάλει ο κύριο Καπέλο, Ιταλική Ιθαγένεια, εξ ονόματο τη Επαρχιακή Ένωση Υπαλλήλων Περιβάλλοντο τη Ιταλία σχετικά με την ε, παρουσία αμοιάντου ε, μεταξύ των ε, σιδηρο, στις σιδηροτροχίες. Ο, αναφέρον δεν είναι πάρα. Και θα δώσω τον λόγο αμέσως στον κύριο Γιάννη Τζιλέκ, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μιλάω εξ ονόματα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και στην παρούσα αναφορά ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι επιβεβαιώθηκαν τα όσα διατηνόταν για την ε, παρουσία μία του μεταξύ συρβιτροχιών και ζητά να γίνει απολύμανση με καθαρισμός ε, προτού συνεχίσει οποιαδήποτε εργασία. αναφέρει ότι η έρευνα η οποία διεξήχθη καταδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων, των εργατών και για οποιοδήποτε, ε, οποιοδήποτε άλλο ε, δουλεύει στις τροχές αυτές. Να επιβεβαιώσω από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι κίνδυνοι αυτοί καλύπτονται από τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα την νομοθεσία οδηγία 2009-148 η οποία προβλέπει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την πρόληψη και την προστασία των εργαζομένων από έκθεση σε αμίαντο και αναφέρει στο άρθρο 3 ότι ισχύει για δραστηριότητες τις οποίες οι εργαζόμενοι, οι εργάτες ε, μπορούν ή ε, εκτίθενται κατά τη δουλειά τους σε υλικά τα οποία ενδέχεται να έχουν αμύαντο, το οποίο ισχύει για την προκειμένη περίπτωση. Η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ αυστηρή, περιλαμβάνει διάφορα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για τους εργάτες, απαγορεύει καταρχάς τις δραστηριότητε που εκθέτουν τους εργάτες ε, σε ίνες αμύαντου ή σε προϊόντα τα οποία έχουν μεταποιημένο μέσα τους αμύαντο. Και σε ό,τι αφορά προϊόντα τα οποία προκύπτουν από κατεδάφιση ε, κτηρίων με αμύαντο. Επίσης, ε, θέτει τα όρια και τις τιμές, ε, τις οριακές για την έκθεση, ορίζει συστήματα και μέσα όπως η παρακολούθηση των κινδύνων, ε, η εκπαίδευση των εργατών και ούτω καθεξής. Του τουλεχθέντος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και αυτή η οδηγία, όπως και άλλες οδηγίες για τις κινδύνους της υγείας, θα πρέπει να μεταφερθούν φυσικά στην εθνική νομοθεσία και ασφαλώς αποκείται στις ε, εθνικές αρχές να εφαρμόζουν στη συνέχεια, στη συνέχεια την νομοθεσία. η νομοθεσία για τον αμύαντο έχει μεταφερθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η περίπτωση που καταγγέλει ο αναφέρον θα πρέπει να καταγγελθεί ενώπιον των Ιταλικών Εθνικών Αρχών έναντι της ε, σχετικής υπηρεσίας επιθεώρησης, η οποία είναι και αρμόδια καταρχάς για τέτοια θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να παρέμβει αν υπήρξε αν υπήρχε ένδειξη παραβίασης εθνικής νομοθεσίας, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αλλά ε, το αντικείμενο της αναφοράς δεν είναι παραβίαση ευρωπαϊκού δικαίου, είναι η ενδεχόμενη επιμόλυνση των συρδιδατροφιών. Και αυτό ε, είναι θέμα αυστηρά εθνικής αρμοδιότητας. Δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό λοιπόν στα γραπτά σχόλια ε, προσθέσαμε τα στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών ε, αρχών της Ιταλίας, της σχετικής επιθεώρησης εργασίας και φυσικά ασφαλώς αν στο μέλλον γίνουν εργασίες ε, καθαρισμού των τροχιών θα πρέπει να συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ειδικότερα με την νομοθεσία, την οδηγία που ανέφερα για τον αμύαντο. Και Φυσικά καλούμε τις Ιταλικές Εθνικές Αρχές να εξετάσουν το θέμα αυτό και αν τυχόν κατά τη φάση της απολύμανσης του καθαρισμού υπάρχουν τεθεί θέμα παραβίασης θα πρέπει να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά επί του παρόντος κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άρα νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναφορά αυτή. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρ θέλει το λόγο. Ναι. Τρεις προτάσεις θα είχα να κάνω. Γιατί και η ίδια η Επιτροπή στην απάντησή της αναφέρει ότι ενδεχομένως να υφίσταται ε, παραβίαση των ελάχιστων προτύπων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας ενδεχομένως. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει το θέμα. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες προς την κατεύθυνση αυτή και θα ήθελα να παραπενθεί το θέμα στην Εθνική Επιτροπή Αναφορών. Γιατί είπατε ότι είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Δεν ξέρουμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει δεν μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση. Εγώ θα παρακαλούσα να γίνει σχετική γνωμοδότηση. Ε, ε, δεν ε, νομίζω ότι υπάρχει τέτοια επιτροπή αναφορών. Υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη που είναι το αντίστοιχο του διαμεσολαβητή, αλλά δεν έχει ακριβώς αυτές τις ε, ε, λειτουργίες. Νομίζω ότι απέναντι σε μια τέτοια καταγγελία, σαν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, σαν Επιτροπή Αναφορών, νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνώσουμε ε, και λίγο διαφορετικά, με πιο ελαστικό τρόπο, την αναφορά αυτή. Δηλαδή δεν μας ζητούν να πάμε να αφαιρέσουμε, από τον αμίαντο από τις ιδιοτροχίες, Απλώς μας ζητούν να παρέμβουμε έτσι ώστε ε, να αποφύγουμε ε, περαιτέρω έργα ε, επί των σιδηροτροχιών αυτών που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε περαιτέρω περιπλοκή της κατάστασης. Εμείς εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ανακοίνωση προς τον αρμόδιο επαλήθευσης ε, της ε, παρουσίας Αμιάντου ε, στην Ιταλία. γιατί αντίθετα από την ε, Εκτελεστική Επιτροπή εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με τους πολίτες έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε λύση των προβλημάτων τους. Επομένως, ε, σαν ε, μια πρώτη φάση μπορούμε να, αφήσουμε, να ενεργοποιήσουμε την αναφορά αυτή και να προχωρήσουμε στις περαιτέρω επαληθεύσεις. Να στείλουμε τώρα, να στείλουμε άμεσα την το να, να αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση απέναντι στις ιδεαλικές αρχές μου φαίνεται ότι δεν είναι της ώρας. Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Ε, είναι, αφορά τη συνέχεια των ε, συζητήσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγού φυσικού αερίου στη Βαλτική θάλασσα του ε, αγωγού, δηλαδή Nord Stream. Δεν είναι παρούσα η συγγήτριά μας. Όμως ζήτησε το λόγο η συνάδελφος Μόρ Μεκνάιτε. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο, η Πρόεδρος, γιατί έχω μάλλον σφαγιάσει το όνομά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κρίμα που δεν είναι εδώ η Δεν μπορώ να μιλήσω επί της ουσίας και του περιεχομένου της έκθεσης, αλλά επειδή ασχολήθηκα με το Nord Stream στο παρελθόν, θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσω τη γνώμη της Επιτροπής για την ε, μελλοντική παρακολούθηση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream. Ε, ξέρω ότι προσφάτως ο θαλάσσιος αγωγός εγκαινιάστηκε με πολύ μεγάλη πολύ θόρυβο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θέματα περιβαλλοντικά και ε, εξάρτησης, ε, ενεργειακής εξάρτησης. Ξέρουμε ότι το Nord Stream όταν έκανε την ε, αξιολόγηση του έργου δημοσίευσε κάποια αποτελέσματα και αποφάνθηκε ότι ο φυσικός αγωγός Nord Stream θα είχε μικρότερο αντίκτυπο, είχε μάλλον μικρότερο αντίκτυπο στον οικότοπο της Βαλτικής από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο να τονίσουμε ότι κάθε χώρα έχει και βλέπει μόνο ένα τμήμα της Βαλτικής. Η τοξικότητα η τοξικότητα. δεν περιλαμβάνεται στην λίστα, στον κατάλογο των παραμέτρων που εξετάστηκαν. Να πω ότι παρά το γεγονός ότι μας ε, χορηγήθηκαν κάποια στοιχεία ε, για την γενετοξικότητα, ε, δεν τονίζεται το ότι έχει αυξηθεί αυτή, ιδιαίτερα για παράδειγμα στην Φιλανδία και σε κάποια άλλα τμήματα της Βαλτικής η γενοτοξικότητα αυτή αυξήθηκε σε εξαπλάσια επίπεδα. και επηρεάζει όλα τα είδη. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι το 2010 δημιουργήθηκε στις ακτογραμμές μία ζώνη υψηλού κινδύνου και η τοξικότητα αυτή εξακολουθεί να αυξάνεται. Φέτος λάβαμε κάποια στοιχεία βάσει των παλιών στατιστικών στοιχείων του 2006-2007 που αναφέρουν ότι μειώνεται το επίπεδο ρήπανση στη Βαλτική. Αλλά όλο όσο ο κόσμος γνωρίζει πόσο κακή είναι η κατάσταση στην Βαλτική και μιλώ και πάλι για την γόνοτοξικότητα και να τονίσω ότι δεν περιλαμβάνουν τέτοια στοιχεία στην έρευνα. Ποια είναι λοιπόν η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Γιατί προγραμματίζεται η, η, η οικοδόμηση τρίτου, τρίτου τμήματος ε, του Nord Stream. Υπάρχουν πληροφορίες οριστικές για το μέλλον και το μελλοντικό αντίκτυπο του Nord Stream στην Βαλτική και στον οικότοπο, θεωρώ ότι η παρακολούθηση των παραβιάσεων αυτών θα πρέπει να δημοσιεύονται. Χρειαζόμαστε επίσης τα τελευταία στατιστικά στοιχεία όταν κάνουμε την σχετική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον αντίκτυπο του Nord Stream, γιατί αυτό δεν τονίζεται επαρκώς. Η Nord Stream αρνείται να χορηγήσει στοιχεία σε ό,τι αφορά την γονοτοξικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να απαιτήσουν τη χορήγηση των στοιχείων αυτών, γιατί από αυτά θα εξαρτηθεί η περαιτέρω επέκταση του Nord Stream. Ε, Ευχαριστώ την συνάδελφο να υπενθυμίσω ότι ε, ε, η βουλευτής ε, είναι εκ των υπογραφώντων την αναφορά. Τώρα είναι βουλευτής, αλλά πριν, πριν γίνει βουλευτής είχε ήδη υπογράψει την αναφορά αυτή. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σας κάνω εξαντλητική ανακοίνωση για το θέμα, γιατί λάβατε το Δεκέμβριο 10 σελίδες για το θέμα, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε πως τα διάφορα θέματα θαλάσσιου, περιβάλλοντος, μεταφορών κτλ. αντιμετωπίστηκαν κατά την διεξαγωγή του έργου αυτού. Πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο έργο και είναι φυσιολογικό να ανακύπτουν σειρά ερωτηματικών σε ό,τι αφορά το θέμα το ενεργειακό, τα θέματα μεταφοράς, θα αναφερθώ σε αυτά που ήδη δήλωσε στη σχετική ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, να εστιαστώ στα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπου θα ήθελα εκ νέου να επαναλάβω ότι το βασικό στοιχείο του ψηφίσματος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή μελέτης αντικτύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι δεν είναι δικό της καθήκον και ότι σύμφωνα με την οδηγία η EIA είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών η διεξαγωγή της μελέτης αντικτύπου. Αυτό και τονίστηκε. Άρα, να επιβεβαιώσω καταρχάς ότι η πρώτη γραμμή έχει ήδη κατασκευαστεί, ότι πρόκειται να κατασκευαστεί σύντομα και η δεύτερη γραμμή και ότι θα ξεκινήσει η διακίνηση αερίου τον Δεκέμβριο και μία από τις απαιτήσει που έχει τεθεί στην Nord Stream από τις τέσσερις ε, χώρες της Βαλτικής και τη Ρωσία είναι ακριβώς η παρακολούθηση της λειτουργίας σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία παρά την, ε, τον περιπλοκό χαρακτήρα της ουσιαστικά αποτελεί ένα σημείο αναφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των καλών πρακτικών, της διαφάνειας που την χαρακτηρίζει. Για παράδειγμα, σε παρόμοια γραμμικά σχέδια, όπως τον Αμπούκο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον χρησιμοποιεί το Nord Stream ως πρότυπο και για άλλα σχετικά σχέδια. Πρόκειται για μια λογιστική προσέγγιση από το α έως το ω αυτή τη σύσταση θα απευθύνει σε όλα τα παρόμοια project η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να επανέλθω τώρα στο συγκεκριμένο θέμα της παρακολούθησης της υποπτίας, να πω ότι διεξάγεται από 20 διαφορετικές εταιρείες μελέτης τις οποίες έχει, με τις οποίες έχει επικοινωνήσει η Nord Stream, όχι μόνο ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά και εθνικά ιδρύματα, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Σουηδικό Εθνικό Μετεωρολογικό και Ιδρολογικό Ίδρυμα. Όλα αυτά τα στοιχεία διορθώνονται, εισάγονται σε μια τράπεζα δεδομένων και χορηγούνται στην ε, χώρα που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση, για την εποπτεία. Για παράδειγμα, στη Γερμανία η βασική υπηρεσία είναι η, το Ιτρογραφικό Ινστιτούτο και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στη Σουηδία, ε, η Σουδιακή Αυτοφυλακή, στη Φιλανδία η σχετική υπηρεσία της ε, Νότιας Φιλανδίας θα σας χορηγήσω τα επακριβή στοιχεία και βάσει αυτής της παρακολούθησης, εάν διαπιστωθούν ε, ανησυχητικά στοιχεία, ε, αναλαμβάνεται δράση. Ως τώρα, σύμφωνα με την μελέτη, με την έρευνα της φιλανδικής αρχή, φιλανδικών αρχών, προκύπτει ότι το έργο δεν έχει παρουσιάσει τόσα προβλήματα όσο αναμενόταν από τον μελέτη δικτύπου. Αντιθέτω, φαίνεται ότι είναι λιγότερα τα προβλήματα από ό,τι αναμενόταν. Συνεχίζεται ωστόσο η παρακολούθηση σε ό,τι αφορά την γενοτοξικότητα. Αυτό το θέμα τονίστηκε από το Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο 6027 κάθετος 2007 και έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν έχουν μεταφραστεί τα έγγραφα αυτά. Ωστόσο, να τονίσω ότι όλες οι σχετικές αρμόδιες αρχές έχουν θεωρήσει ότι δεν είναι τέτοιο επίπεδου η γονιδιακή τοξικότητα ώστε να χρειάζονται ανάληψη δράσης. αυτό το θέμα της ε, τοξικότητας αυτής δεν ε, τέθηκε κατά την τριετή περίοδο εξέταση της μελέτης αντικτύπου. Φυσικά μπορεί να πρόκειται για ένα νέο στοιχείο, ωστόσο θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των υποχρεώσεων των κρατών ε, μελών στα πλαίσια της οδηγίας για το θαλάσσιο περιβάλλον και των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Nord Stream. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για τη βαλτική και για την γονιδιακή τοξικότητα και όταν τα στοιχεία αυτά θα τα έχουμε στην διάθεσή μας, ασφαλώς και θα σας τα διαβιβάσουμε. Όχι μόνο σε εσά, στους βουλευτές, αλλά σε όλους. Άρα, κλείνοντας από πλευράς περιβαλλοντικής προστασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι υπήρξε παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Αντιθέτω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη έχουν κερδίσει πολύτιμες εμπειρίε από την εμπειρία του Nord Stream και θα θέλαμε να τη μοιραστούμε την εμπειρία αυτή με άλλα προγράμματα μέσω ενός σχετικού εγγράφου. Και για τα υπόλοιπα σας παραπέμπω στην ανακοίνωση που δημοσίευσαμε. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, απάντηση. Οπωσδήποτε θα μας ξανααπασχολήσει το θέμα ε, στο μέλλον. Ελπίζω ε, την παρουσία της εισηγετρίας έτσι ώστε να αποφασίσουμε ποια θα είναι η συνέχεια που θα δώσουμε στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο που υπέβαλε την αναφορά αυτή. Περνάω στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Είναι η αναφορά του κυρίου Άσπροκ εξ ονόματος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Εργαζομένων Αλληλεγγύη Ανεξαρτησία Δημοκρατία ΣΥΝΤ ε, που υποστηρίζεται και από άλλες 469 υπογραφές. Ο αναφέρον ε, θεωρητικός πρέπει να είναι μεταξύ μας. Ναι, ναι, και θα δώσω αμέσως ε, τον λόγο. Πρόεδρε, φίλοι Ευρωπαίοι, Κύριε Βαλέσα, μακάρι να είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Συμβασιούχο και τον κύριο κύριο έκτακτο. Ο ένας περνάει ένα διαγωνισμό και παίρνει ε, δουλειά ως συμβασίουχος. Δεν του επιτρέπεται να συμμετέχει στις ιστορικούς διαγωνισμούς. Και ύστερα έχουμε τον κύριο Έκτατο, ο οποίος ζητά δουλειά ω έκτακτος υπάλληλο. Του μιλάνε λίγο, του δίνει, τους δίνει και το βιογραφικό τους και παίρνει τη δουλειά και έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Επιτροπή σε ιστορικούς διαγωνισμούς. Και ο λόγος γιατί είναι σημαντικό αυτό είναι ο εξής. Στους ιστορικούς διαγωνισμούς το ποσοστό επιτυχίας το παραδέχεται ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 25%. Ένα στα τέσσερα. Να πάρεις μια δουλειά για την υπόλοιπη ζωή σου. Στους εξωτερικούς διαγωνισμούς που πέρασα και εγώ για παράδειγμα είναι 1% στην καλύτερη περίπτωση, ένα στους χίλιους στην χειρότερη. Τι ζητάμε. Να έχουν τα ίδια δικαιώματα οι έκτακτοι με τους σημασιούχους. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος, ούτε θεατολογικός ούτε νομοθετικός για να γίνεται η διάκριση αυτή και να σας υπενθυμίσω σύντομα την αστεία αλλά ενοχλητική περίπτωση του Βαρόνου Φον Γκουτουμπέρκ στην Γερμανία, όπου ανακαλύψαμε ότι το PhD του, το διδακτορικό του, ήταν κλεμμένο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτό παραβιάζει τα δικαιώματα υπό το χάρτη των, ανθρωπινών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των εκτακτών συμμεσίουχων υπαλλήλων. Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε τέτοια. Και την ε, οδηγία 1999 ε, κάθετος 70 ε, Και θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό που ζητάμε θα είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή αλλά απτή εξοικονόμηση. Και γιατί, γιατί όσο πιο πολλοί κόσμος έχει πρόσβαση στους ιστορικούς διαγωνισμούς, τόσο πιο υψηλό θα είναι το επίπεδο του μέσου επιτυχόντος. Άρα, το να ανοίξει η διαδικασία αυτή και στους έκτακτους υπαλλήλους θα βελτιώσει τη ε, ποιότητα των υπαλλήλων μας κατά 1% έστω. Και να θυμάστε ότι μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν ήδη δώσει τα βιογραφικά τους, έχουν περάσει ήδη έναν διαγωνισμό και άτομα τα οποία έχουν ήδη έχουν εργαστεί επί σειρά ετών στην Επιτροπή. Άρα θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ πρακτική σύσταση. Αν τώρα στη συνέχεια κάποιος έχει, έχει κάνει ερωτήσεις, ε, ευχαρίστως να απαντήσω στα αγγλικά, στα γαλλικά ή και στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας παρακαλώ βοηθήστε μας να δώσουμε στους συμβασιούχους τα πλήρη τους δικαιώματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέγομαι Ρομπέρτο Καρλίνη και είμαι υπεύθυνο ε, της ε, διεύθυνσης ε, concorsi presso la nostra προσλήψεων ε, στην ε, Γενική Διεύθυνση Προσωπικού. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε δύο-τρία στοιχεία απαντώντας στα όσα είπε ο κύριος Άσπρουκ ε, εξ ονόματος του Ιδίου και των υπολείπων αναφερόντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει μια γραπτή απάντηση στην Επιτροπή σας το 2009 όπου αναφέρονται ε, και μελετώνται λεπτομερία τα τρία στοιχεία της αναφοράς. Το πρώτο το οποίο αφορούσε τον αποκλεισμό συναδέλφων που είναι ταυτόχρονα ε, και πολίτες ε, των 15 πρώτων χωρών αυτό αναλύθηκε ε, και ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά ε, τις ε, προσλήψεις ε, δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν εξαιρέσεις για τις χώρες της διεύρυνσης των 10 και τις χώρες της διεύρυνσης των 2 και επίσης αναφέρεται και στο άρθρο 2 του καταστατικού που λέει ότι θα πρέπει να προσαρμόζεται η γεωγραφική κατανομή όσο γίνεται πιο γρήγορα στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημείο το οποίο έθιξε και σήμερα ο κύριος Άσπροκ αφορά το γεγονό ότι αυτοί οι εσωτερικοί κανονισμοί θα έπρεπε να ε, είναι ανοιχτοί ε, και ε, στους συμβασιούχους και όχι μόνο στους μόνιμους και τους έκτακτους υπαλλήλου. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 29 όπου δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια και εάν ε, ε, πραγματικά θέλουμε να κατανοήσουμε την, ε, το, το πνεύμα του νομοθέτη, θα πρέπει να δούμε ότι στο οργανόγραμμα δεν καλύπτονται μονάχα οι θέσεις των μονίμων και των εκτάκτων. Οι συμβασιούχοι όσον αφορά το καταστατικό ε, του προϋπολογισμού δεν αναφέρονται ε, στο οργανόγραμμα αλλά σε κάποιους ε, ειδικού καταλόγους. Υπάρχουν λοιπόν θέσεις τις οποίες ήδη καλύπτουν κάποιοι έκτακτοι υπάλληλοι και όταν γίνουν μόνιμοι περνώντας το διαγωνισμό μπορούν πλέον ως μόνιμοι να καταλάβουν την ίδια θέση. Τρίτο, στοιχείο ε, και είναι ε, αυτό το οποίο αφορά την, το κατά πόσο είναι απλή η διαγωνισμή αυτή. Ε, γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διαγωνισμοί της διεύρυνσης των 10 που ακολουθήθηκαν σε μια δεύτερη φάση από τις, χώρες, τις δύο χώρες της τελευταίας διεύρυνσης ε, ήταν κάπως ειδική. Ε, κατανοούμε ότι ε, έπρεπε να δοθεί μία απάντηση στην μεγάλη ανάγκη προσωπικού και για να απαντήσω όμως στην κατηγορία της, των υπερβολικά απλών διαγωνισμών πρέπει να πω ότι οι διαγωνισμοί αυτοί οργανώθηκαν με τη συμβολή της ΕΠΣΟ. και η, τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Άσπροκ όσον αφορά ε, την, ε, το ποσοστό επιτυχίας ε, είναι κάπως υπερεκτιμημένη. Εμείς λέμε ότι είχαμε ποσοστό επιτυχίας 23% για τους ε15 και 26% για τους ε2 όσον αφορά τις προσλήψεις, γιατί βεβαίως πρέπει να δούμε πόσοι είναι αυτοί που πραγματικά προσελήφθησαν από τους καταλόγους των επιτυχόντων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό πρόσληψης σε σχέση με τις θέσεις που ήταν ε, που είχαμε διαθέσιμες για τις ε12 ε και ε12 ε, που έχει φτάσει στο ποσοστό 16%. Ε, σε ε, σύνολο λοιπόν 4.000 και κάτι ε12 και ε2 έχουμε μονάχα ένα ποσοστό 12% τελικής επιτυχίας οι άλλοι συνάδελφοι προσελήφθησαν μέσω γενικών διαγωνισμών ε10 ε, και ε2 ε, ε, με την συνδρομή της ΕΠΣΟ και βεβαίως υπήρξαν και οι αιτήσιοι διαγωνισμοί της ΕΠΣΟ όπου, που είναι ανοιχτοί και που μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Νομίζω ότι αυτά ε, τα στοιχεία είναι αρκετά για την ώρα και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ σας. Ευχαριστώ πολύ κύριο Καρλίνη. Ο κύριος Γιάννη έχει το λόγο. Να κάνω την εξή πρόταση επειδή έχει περάσει και η ώρα. Σε ό,τι αφορά την ε, ύπαρξη μη διακριτικής μεταχείρισης. Είναι νομικό το ζήτημα. Ο... Η Επιτροπή αναφέρεται στο καταστατικό για τις προσλήψεις. Κατά πόσον ε, πληρούνται οι μη οι όροι για την διακριτική μεταχείριση. Θα προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να μεταφερθεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες. Να μεταβιβαστεί, να αναπαφευθεί η αναφορά στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και η οποία και να γνωμοδοτήσει για να αποφασίσει η σχετική λοιπόν Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Αυτή θα ήταν η πρότασή μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και νομίζω ότι συμμερίζομαι την πρόταση του Γιάρ, δηλαδή θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θα ζητήσουμε γνωμοδότηση από την Γιούρη σε σχέση με το θέμα που έθιξε ο αναφέρον. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη, η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.